Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, α αρχίσουμε γιατί έχουμε πολλά πράγματα στην ημερήσια διάταξη και θέλω να σα καλωσορίσω όσοι είσαστε ήδη εδώ και κυρίω έτσι την έναρξη τη συνεδρίασης. Όσοι ήθιστε να ξέρετε ότι μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίασή μα όπω πάντα και το πρώτο θέμα που έχουμε είναι η έγκριση τη ημερήσιας διάταξη. Την πήρατε στι 4 Οκτωβρίου την τελική μας ημερήσια διάταξη, μία αλλαγή έχουμε μετά από έτοιμα του ΕΛΚ και στηρίζουν και οι σοσιαλιστές ε, και οι άλλοι να αναβληθεί η ψηφοφορία της έκθεσης του Ρίτσαρτ Κόρμπετ που είναι το σημείο 9 στην ημερήσια διάταξη. Και αυτό γιατί πρέπει να συνεχιστούν οι συζητήσεις για τις συμβαστικές τροπολογίες και δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Οπότε εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη με αυτή την τροποποίηση. Το δεύτερο που έχω να σας πω στις ανακοινώσεις μου, πρώτα απ' όλα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στους προπολογισμού για το 2019. Η Επιτροπή Προπολογισμών λοιπόν ψήφισε την θέση της ως προς το Συμβούλιο για τον προπολογισμό αυτό και οι παρατηρήσεις της ΑΦΚΟ, κάποιες εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Προπολογισμών κάποιες τροπολογίες ε, για την ανακοίνωση της ε, Κομισιόν όσον αφορά τον διάλογο των ε, πολιτών, το European Public Spaces και το Europe for Citizens. Για αυτές τις δύο τελευταίες εμείς ζητούσαμε να επανέλθει η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα ποσά, αλλά το Συμβούλιο τελικά δεν έκανε περικοπές, οπότε ήταν περιττό να ψηφιστούν, γιατί δεν έγιναν περικοπές και δεν χρειαζόταν να επανέλθουν τα ποσά. Οπότε είμαστε στη γραμμή που θέλαμε. Και μετά υπάρχει ένα θέμα που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Είχαμε επιλοτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν μη εφαρμόσιμα οι τροποποίησεις μας αυτές. Υπήρξε μεγάλη μείωση όσον αφορά την ε, στήριξη λοιπόν. Ε, η Επιτροπή αποφάσισε ότι δεν είναι εφαρμόσιμο, οπότε δεν τέθηκαν και σε ψηφοφορία. Μπορούμε βέβαια φυσικά πάντα να έχουμε από μεμονωμένους βουλευτές ε, επανυποβολή των τροπολογιών αυτών, αλλά η πιθανότητα να εγκριθούν είναι πάρα πολύ μικρή. Γιατί τα ποσά δεν επιτρέπουν καμία μετακίνηση. Οπότε δεν θα μπορέσουν να συμπεριληφθούν, πιστεύω. Η θεωρητικά όμως η δυνατότητα υπάρχει να τις υποβάλλετε και πάλι. Και εφόσον το θέλετε, η γραμματεία είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει. Ο Ζωζέ μου λέει ότι θα έπρεπε να αποφασίσουμε καλύτερα εάν θα προβούμε σε αυτήν την επανυποβολή ή όχι. Να ξέρουμε, ξέροντα βέβαια πάντα ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πετύχουμε, δεν θα περάσουν. Αλλά αν εσεί αποφασίσετε να το κάνουμε, πείτε μου, θέλετε, όχι, παρετούμαστε από αυτέ. Ωραία, καλώ. Τώρα και πάλι, βέβαια κάποιοι λείπουν, αλλά πρόσφατα ε, διάφοροι από εσά διαμαρτυρηθήκατε ότι έχουμε πάρα πολλέ συναντήσει, για παράδειγμα στο Στρασβούργο, τις Δευτέρες το βράδυ, αλλά αυτό έχει να κάνει με την απόφαση που εμείς ήδη πήραμε για τις εκθέσεις που θέλαμε να εκπονήσουμε, τις νομοδοτήσεις και είναι και απόφαση του διάσκεψης των Προέδρων που έχει βάλει προθεσμία για την ψηφοφορία στις κοινοβουλευτικές επιτροπές όσον αφορά τις εκθέσεις πρωτοβουλίας που μπορούν να ψηφιστούν το αργότερο μέχρι τις 27 Νοεμβρίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο πρέπει να ολοκληρώσουμε το έργο μας για τις εκθέσεις πρωτοβουλίας. Γι' αυτό και έχουμε όσες ε, συνεδριάσεις χρειάζεται να έχουμε και όσο περισσότερο έχετε τόσο το καλύτερο. Δεν μπορώ να μειώσω τον αριθμό των ε, συνεδριάσεων και δεν μπορώ να μειώσω το έργο που πρέπει να επιτελέσουμε. Έτσι είναι όμως. Και είναι κάτι που έχουμε αποφασίσει από κοινού. δύο φορές το εξήγησα. Έχουμε μεγάλο φόρτο εργασίας, αλλά θα συνεχίσουμε. Μετά θα έρθει και η διαδικασία της σύμφωνης γνώμης και θα έχουμε άλλες συνεδρίσεις γι' αυτό. Κάτι άλλο τώρα, πάντα στις ανακοινώσεις μου. Αποφάσεις των συντονιστών με τη γραπτή διαδικασία. Δεν είχαμε χρόνο την προηγούμενη εβδομάδα για να αποφασίσουμε διαφορετικά. Όσον αφορά τις αποστολές λοιπόν, πρώτα απ' όλα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο τη σύστησαν την αποστολή αυτή και μπορεί να γίνει την εβδομάδα 9, 28 Φεβρουαρίου με 1 Μαρτίου. Μόνο τις λεγόμενες πράσινες ημέρες μπορούμε, όπως ξέρετε, και είναι οι μόνες που έχουμε το πρώτο ήμιση του 2019. Ήταν η μόνη δυνατότητα που είχαμε από τον Ιανουάριο μέχρι το τέλος της θητείας μας. Υπάρχει και σύσταση επίσης από τους συντονιστές να συναντηθούμε και πάλι με εκπροσώπους της Επιτροπής της Βενετίας. Θα θυμόσαστε ότι είχαμε ήδη μία πολύ καλή, αλλά θα μπορούσαμε να το ξανακάνουμε στο Στρασβούργο, ίσως σε κάποια ολομέλεια στο Στρασβούργο. Και εφόσον γίνει έτσι δεν χρειάζεται καν άδεια για ποσόστοση όσον αφορά ταξίδια κτλ. Αυτό όσον αφορά τις αποστολές. Μία θα πάμε και μία άλλη θα έρθουν εκπρόσωποι της Επιτροπής της Βενετίας στο Στρασβούρο. Για τις ακροάσεις τώρα. Τρεις σύστησαν και συμφώνησαν οι συντονιστές μέσω της γραπτής διαδικασίας. Η πρώτη ακρόαση θα θυμόσαστε ότι είχαμε συζητήσει για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όσον αφορά την επικοινωνία με τον κόσμο και μάλιστα εν ώψη των εκλογών. Οπότε υπάρχει μια ακρόαση που προβλέπεται λοιπόν για τις ευρωπαϊκές κοινοβουλευτικές εκλογές, ευρωπαϊκά κόμματα και ευρωπαίοι ψηφοφόροι. Αυτή θα είναι μια ακρόαση. Η δεύτερη είναι πρόταση που πολύ πιθανόν ε, να καταλήξει σε κοινή οργάνωση ακρόασης με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Έχει να κάνει με τη συνταγματική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την συνταγματική δράση και αντίδραση μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης. Αυτή είναι η πρόταση που στήριξαν οι συντονιστές. Και η τρίτη προβλεπόμενη ακρόαση είναι ότι μπορούμε να οργανώσουμε μια ακρόαση για τις επιμερισμένες αρμοδιότητες, εκτελεστικές αρμοδιότητες, επιμερισμένες μεταξύ κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με παραδείγματα από την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή. Και αυτή η ακρόαση θα διεξαχθεί από κοινού με την ΛΥΜΠΕ, σε συνεργασία με την Επιτροπή Λευθεριών του Πολίτη. Συνεπώς πρέπει να ελέγξουμε με την ΑΦΕΤ και τη ΛΥΜΠΕ, να δούμε αν συμφωνούν ώστε οι δύο τελευταίε ακροασει να οργανωθούν από κοινού. Αντιρρήσει. όχι από ό,τι βλέπω, οπότε θεωρώ ότι η Επιτροπή μα εγκρίνει τις αποφάσεις αυτές των συντονιστών. Τρίτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, έγκριση των πρακτικών. Πρόκειται για τη συνεδρίασή μας 26 και 27 Φεβρουαρίου. Τα πρακτικά είναι στη διάθεσή σας και σύμφωνα με την συνήθη πρακτική μας, αν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, τότε θεωρούνται εγκεκριμένα τα πρακτικά αυτά. Επίσης, να σας πω λίγο σύντομα τι έγινε από την προηγούμενη Δευτέρα μέχρι σήμερα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το Brexit, την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Είχα δύο διμερείς συναντήσεις αυτές τις δύο τελευταίες εβδομάδες με τον μόνιμο εκπρόσωπο του, το... κάτω χωρών, τον Ρόμπερ Ντεχρότ, ο οποίος με ενημέρωσε, και σας το λέω και εγώ, για την προετοιμασία που γίνεται σε επίπεδο χωρών μελών, σε διάφορα διοικητικά επίπεδα. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τεράστιο έργο. Για μερικές χώρες μάλιστα είναι πολύ μεγαλύτερη πρόκληση από ό,τι για άλλες. Οι κατοχώρες έχουν πάρα πολλά λιμάνια, για παράδειγμα, που είναι πολύ σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν ένα θέμα. Και βέβαια συζητήσαμε και για την ενότητα μεταξύ των χωρών μελών και τις κόκκινες γραμμές που έχουν υιοθετηθεί μέχρι τώρα από εμά για τις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή δεν παρετούμεθα από την ενιαγορά, για παράδειγμα ένα πολύ βασικό. Και μετά συναντήθηκα και με τον Ιρλανδό Υπουργό για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, την κυρία Έλεν Μακεντή. Ε, και συζητήσαμε μαζί για νομικά ζητήματα, θέματα συνόρων, ειρηνευτική διαδικασία, πώς θα την προστατεύσουμε. Και επιβεβαιώθηκε η δέσμευση της Ιρλανδίας υπέρ μιας ε, λύσης για το Ιρλανδικό να μπορέσουμε να καταλήξουμε δηλαδή κάπου με τις διαπραγματεύσεις αυτές. Ε, σήμερα έχουμε και το steering group. Από όσο ξέρω, συνεχίζονται οι τεχνικού χαρακτήρα ε, διαπραγματεύσεις, όχι πολιτικού τύπου αυτή τη βδομάδα. Και τώρα έχουμε λίγο χρόνο πια για να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις. Θυμόσαστε ότι είχαμε δεσμευτεί ότι στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου που έχει ένα δείπνο σε μια εβδομάδα για το Brexit, εκεί πρέπει να υπάρξει δυνατότητα για τον Μισελ Μπαρνιέ να πει ότι υπάρχει αποφασιστική σημασίας πρόοδος ώστε να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποφασίσει στη συνέχεια για το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα είναι νομίζω την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου. Και εκεί να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Και στη συνέχεια, μετά από μερικές εβδομάδες, το Συμβούλιο θα μπορεί να στείλει την συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μετά θα μπούμε στην επίσημη τυπική διαδικασία. Θα σας πω το δικό μου προσωπικό σχόλιο. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να διαρρεύσουν κάποια πράγματα από τη συμφωνία. Αλλά έτσι κι αλλιώ, αν διαβάσετε τα μέσα ενημέρωση, τι λένε. Πάνε πάνω κάτω. Δηλαδή, μια μέρα λένε δεν υπάρχει συμφωνία, την άλλη μέρα λένε ότι φτάνουμε σε συμφωνία. Πρέπει να περιμένουμε. Έχουμε κάποιες μέρες πριν από το δείπνο της Τετάρτης και από τον Μισελ θα πρέπει να ακούσουμε όχι ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσει, αλλά ότι υπάρχει αποφασιστική σημασία πρόοδο και μετά θα δούμε τι θα γίνει και με τις πολιτικές δηλώσεις. Αυτά νομίζω είχα να σας πω. Μην ξεχνάμε ότι την 1η ε, Απριλίου, εφόσον όλα πάνε καλά, θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον, τη μελλοντική σχέση. Και εκεί πρέπει να υπάρχει εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ ξέρετε ότι γίνονται πολλές προετοιμασίες, σεμινάρια κτλ. στην Κομισιόν, αλλά είναι πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε γι' αυτό και να αποφασίσουμε. Και όσον αφορά την προετοιμασία πρέπει να σας πω, γιατί περιμένουμε κάποια στιγμή πριν τα τέλη της χρονιάς, θα ακούσουμε από την Επιτροπή τι προτάσεις έχει στην περίπτωση μη συμφωνίας. Τι θα έχει να προτείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κομισιόν. Ακούσαμε ήδη για το χρηματοπιστωτικό κλάδο, αν δεν υπάρξει συμφωνία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, περιμένουμε ανακοίνωση για προτάσεις σε περίπτωση μη συμφωνίας, ανάλογα βέβαια με το πώς θα προχωρήσουν και οι διαπραγματεύσεις, αν θα έχει υπάρξει αποφασιστική σημασία πρόοδος ή όχι. Ρίτσαρτ, για το Brexit τελείωσα. Θα περούσα στο σημείο 5, αλλά αν έχει κάτι να σχολιάσεις, παρακαλώ. Πες. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά αυτά που είπες για την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας. Υπάρχει και δυνατότητα, που εγώ λέω ότι είναι ο κίνδυνος, να υπάρξει μια συμφωνία που δεν θα λέει τίποτα, που θα αναβάλει όλα τα σημαντικά στοιχεία για μετά το Brexit. Αυτό κάποιοι το λένε μια, ένα τυφλό Brexit, δηλαδή που θα μένουν όλα τα ζητήματα για το μέλλον και δεν θα έχει λυθεί τίποτα. Η δήλωση για την μελλοντική σχέση μπορεί να περιλαμβάνει μόνο γενικότητες και να μην δίνει καθόλου ενδείξεις για το πώς θα λυθούν τα διάφορα ζητήματα. Αν όντω είναι έτσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Βρετανικό Κοινοβούλιο θα κληθούμε να ακυρώσουμε τη Συμφωνία Αποχώρησης χωρίς να έχει λυθεί κανένα στοιχείο κλειδί, χωρίς να γνωρίζουμε δηλαδή που πάμε στο μέλλον. Και εγώ κάνω έκκληση σε όσους συμμετέχουν στις συζητήσεις να φροντίσουν να μην καταλήξουμε σε κάτι τέτοιο, γιατί δημοκρατικά είναι απαράδεκτο. Και διαδικαστικά και για το μελλοντικό σχεδιασμό δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Έχω και ένα δεύτερο σημείο. Είπατε ότι τον Νοέμβριο μπορεί να υπάρξει κάτι που παραπέμπει στη συμφωνία και θα αρχίσουμε τις διαδικασίες για να υπάρξει σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά πάσα πιθανότητα στην πρώτη ολομέλεια του Μαρτίου. Μπορεί να υπάρχει και ένα πρώτο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άπαξ και ανακοινωθεί ότι υπάρχει συμφωνία, σαν μια πρώτη αντίδραση και ίσως να λέμε θέλουμε περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό, θέλουμε μεγαλύτερη δέσμευση για το άλλο και ίσως να μπορούμε να πούμε ότι και το ένα ή το άλλο ζήτημα τα θεωρούμε απαράδεκτα και ότι θα έπρεπε να ξαναμπούν σε διαπραγμάτευση. Ε, η διευθύνουσα ομάδα, το steering group, νομίζω ότι το έχει συζητήσει. Ισχύει, μπορεί να γίνει αυτό ή έχει εγκαταληφθεί αυτή η ιδέα. Μαρτίν Άντερσον. Ευχαριστώ και εγώ. Μια που περιμένουμε τώρα το κείμενο της Βρετανικής κυβέρνησης για τη δικιά τους εκδοχή της ε, νομικής δέσμευσης που αναλαμβάνουν, να ξέρετε ότι διαβάσαμε για 75% αυτό που θέλανε 75% των ε, συντηρητικών δηλαδή και φαίνεται ότι είναι αρκετά επικίνδυνο. Δεν είναι έτσι. Έλεγα λοιπόν ότι είμαστε εν αναμονή του κειμένου της Βρετανικής κυβέρνησης για το πρωτόκολλο, το νομικά δεσμευτικό, τη δικιά του εκδοχή δηλαδή για την κατάσταση στην Ιρλανδία. Και είναι ανησυχητικό που ακούμε ότι 75% των συντηρητικών είπαν ότι είναι διατεθειμένοι να παραιτηθούν από την συμφωνία με την Ιρλανδία προκειμένου να πετύχουν το Brexit. Καταλαβαίνετε ότι αυτά που τα ακούμε εμεί στην Ιρλανδία είναι κάτι τρομερό και αδίσταχτο. Με τόση δουλειά που έχει κάνει η Επιτροπή μας για την διαδικασία Ο Μισελονίλ ήταν ε, την ε, Παρασκευή με την αντιπροσωπή εδώ ως αντιπρόεδρος ε, του Sinn με τον Κολιούτσχουτ, με τους Πράσινους και με το κόμμα της Συμμαχίας και όλοι, όλα τα κόμματα στηρίζουν και η πλειοψηφία του κόσμου στη Βόρεια Ιρλανδία και είναι κατά κάτι τέτοιο. Το παράρτημα 1 που δημοσιεύτηκε για τα δικαιώματα. Υπάρχει μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων για δικαιοσύνη κλπ. που έχει προσφύγει στην υπηρεσία της Ευρωπαίας Ombudsman ακριβώς επειδή ανησυχούν για τα θέματα δικαίου και δικαιωμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα και το οποίο συμφώνησε η Βρετανική κυβέρνηση το Δεκέμβριο και που δεν προσφέρει αρκετές εγγύσεις. Λοιπόν, για αυτά που είπε ο Ρίτσαρτ, για την ε, δυνατότητα να μην ε, προχωρήσουμε, η υπάρχει ανησυχία από την πλειοψηφία, την πλειοψηφία του κόσμου κλπ. Στηρίζουμε το backstop να ενισχυθεί και όχι αυτά που ακούμε από την Βρετανική κυβέρνηση και που μας ανησυχούν. Η νοτροπία η αγγλική φαίνεται ότι προσπαθούν να την ε, προχωρήσουν και να την καθετρήσουν στο βορρά μέσω ενό κόμματο που δεν είναι όμω η πλειοψηφία του κόσμου και δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τον κόσμο της Βόρειας Ιλανδίας. Ο κόσμος αρχίζει να ανησυχεί για την ιδέα αυτή του πραγματικού συνόρου στην Ιρλανδία. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή η διευκόλυνση υπάρχει χρόνια στην Ιρλανδική θάλασσα. Οι υπάλληλοι στο βορρά, που είναι ουδέτεροι σε σχέση με τα πολιτικά κόμματα, έχουν υποβάλει πρόταση για την διευκόλυνση αυτή να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να μην γίνει ε, περισσότερο σκληρό, όπως λέμε, το σύνορο, τα σύνορα στην Ιρλανδία. Πρέπει να στηριχτεί η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, όπως θέλει ο κόσμος στη Βόρεια Ιρλανδία. Όλα πρέπει να τηρηθούν και η Βρετανική κυβέρνηση πρέπει να τα σέβεται. Δεν πρέπει να βρουν μια διατύπωση που θα αποδυναμώνει αυτή τη συμφωνία. Μια συμφωνία την οποία έχει στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι χώρες που είναι υπέρ της ειρήνης και που έχει και κόκκινες γραμμές. Έχουμε πει ότι θα τηρηθεί πλήρως. Δεν πρέπει να υπάρξουν αυτά τα σύνορα. Εμείς καταδικάζουμε την οτροπία αυτών που είπαν επίσης ότι θα αφήσουν να καταρρεύσει η ειρήνη προκειμένου να πετύχει το Brexit όπως το θέλουν. Δεν μπορεί να είναι αυτή η θέση κανενός και αυτό πρέπει να το καταδικάσουμε. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλε ανακοινώσει στην ανακοίνωση μου. Να σα πω τι είπα, τι άκουσα μάλλον. Την περασμένη εβδομάδα σαν διευθύνουσα ομάδα για το Brexit, εκδώσαμε μια δήλωση. Αφορούσε την ανάγκη τατικοποίησης των διαπραγματεύσεων. Να έχουμε αποφασιστική πρόοδο εγκαίρω. Να μειωθεί ο κίνδυνος ελλείψεω συμφωνίας. Τώρα, αν θα υπάρξει άλλο ψήφισμα δεν ξέρω. Αρχικά είχαμε πει ότι ίσως τον Οκτώβριο να έχουμε άλλο ένα για την Ιθαγένεια. Άλλο ένα ψήφισμα. Δεν το επεξεργαζόμαστε ακόμα, θα σας ενημερώσω αν καταλήξουμε σε αυτό. Τώρα, όσον αφορά τη διαδικασία σύμφωνης γνώμης, το ξέρετε καλύτερα από μένα, λόγω της δουλειάς που κάνετε τελευταία χρόνια, για τον εσωτερικό κανονισμό που χρησιμοποιήσουμε το άρθρο 99 και να έχουμε ένα ψήφισμα που θα συνοδεύει το κείμενο τη Συμφώνου Γνώμης Επιτροπής. Μπορεί να υπάρχει και άλλη μια απόφαση για ξεχωριστή ε, ξεχωριστό ψήφισμα των πολιτικών ομάδων νωρίτερα που δεν θα σχετίζεται με τη διαδικασία συμφώνου γνώμη. Δεν έχω ακόμα κάποιες ειδήσει. Θα πρέπει να αποφασίσουμε τη δεδομένη στιγμή. Τι θα κάνουμε. Και όσον αφορά το περιεχόμενο πολιτικής δήλωσης, θα, θα θυμάσαι, Ρίτσαρντ, ότι άλλαξε κάπως η διάθεση τον τελευταίο χρόνο. θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να είναι πολύ γενικόλογη δήλωση. Μετά μπήκαμε σε λεπτομερέστατη δήλωση και τώρα η προσέγγιση είναι πιο ισορροπημένη. Θα πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερής, το ώστε να μπορούμε να δούμε και εμείς το περιεχόμενο και να μπορεί και η Βρετανική πλευρά να ψηφίσει θετικά. Για να το κάνει αυτό, πρέπει να έχει σαφείς κατευθύνσεις για το μέλλον. Δεν ξέρω ποια θα είναι τελική πολιτική δήλωση. Είναι σαφέ το κείμενο δεν μπορεί να είναι νομικά δεσμευτικό. Θα είναι πολιτική φύσεω η δήλωση. Αν θα σχετίζεται τώρα με τη συμφωνία απόσυρση ή όχι, δύσκολο να το πω. Και εκεί έχουμε εξελίξει. Τώρα τελευταία κατάλαβα ότι έγινε λιγότερο σημαντικό για τους Βρετανούς να υπάρχει σαφής διασύνδεση. Μπορεί να ολοκληρωθεί η συμφωνία απόσυρση και ολοκληρωθεί η πριν τη Σύνοδο Κορυφή του Οκτωβρίου και μετά να αρχίσουν οι εργασίες στην πολιτική δήλωση. Ο Μισελ Μπαρνιέ είπε ότι όλα αυτά τα πράγματα που σχετίζονται με εξωτερική ασφάλεια και εξωτερική πολιτική ε, ήταν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Άρα έχει εξασφαλιστεί ένα τμήμα της πολιτικής δηλώσεως. Έχει εξασφαλιστεί ότι θα συμπεριληφθεί σαν θέμα και πολλά μέτρα και εργαλεία στηρίζονται από τις δύο πλευρές για την εσωτερική ασφάλεια Ίσως δεν υπήρξε τέτοιο βαθμό συμφωνία για τις θελικέ προτάσεις, αλλά φαίνεται ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Εκκρεμότητα είναι το οικονομικό τμήμα. Τώρα, αν θα είναι αρκετά λεπτό μέσα στο κείμενο, θα δούμε. Αλλά υπάρχει συνεννόηση, κατανόηση πλευρά Μπαρνιέ ότι δεν θα απεψηφίσουμε για μια πολιτική δήλωση κενή περιεχομένου. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δει κάποιες δεσμεύσεις. Δεν θα είναι δεσμευτικό όμως, γιατί πολύ συχνά από του Βρετανούς ακούσαμε ότι η μελλοντική κυβέρνηση μπορεί να αγνοήσει τα πάντα. Πρέπει να πετύχουμε την ισορροπία μεταξύ λεπτομερία που μπορεί να συμπεριληφθεί και γενικόλογη προσέγγιση. όπως συνήθω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το γενικόλογο κείμενο επιτρέπει ευελιξία για διαπραγματεύσει. Να πω και κάτι άλλο. Α, έφυγε η Μαρτίνα. Η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πάντα ότι για το Ιρλανδικό ζήτημα είχαμε ένα όριο, ένα backstop. Πιστεύαμε ότι δεν υπονομεύεται η συνταγματική ακαιρεότητα του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά ήμασταν ανοιχτοί σε οτιδήποτε θα προχώταν από τη Βρετανική πλευρά για να βελτιώσουμε αυτό το μέτρο, το backstop και αυτό έγινε στις πρόσφατες ε, διαπραγματεύσεις. Έχουμε δέσμευση για προάσπιση συμφωνίας Μεγάλης Παρασκευής της συνευτικής διαδικασίας. Ε, Ήταν και η κόκκινη γραμμή που είχαμε θέσει από την αρχή. Πρέπει να την κρατήσουμε. Δεν ξέρω τι θα προτείνει το Ενωμένο Βασίλειο τις επόμενες ημέρες. Αυτά εν είδη σχολείου. Πάμε παρακάτω. Μπάρμπαρα Σπινέλη. Εφαρμογή της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη διεξήχθησαν κάποιες συζητήσεις, Μπάρμπαρα. Συμφώνησες να είσαι όσο πιο λακωνική γίνεται για να ολοκληρωθεί η εξέταση σήμερα του εγγράφου εργασίας. Έχει το λόγο, Μπάρμπαρα. Ευχαριστώ, Ντανούτα. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνέβαλαν στην παραγωγή του εγγράφου εργασίας και τους εμπειρογνώμονες εξωτερικούς που συμμετείχαν στη φάση των ερευνών και τους συναδέλφους του Κοινοβουλίου και τους διάφορους εκπροσώπους του προσωπικού που συμμετείχαν στις διάφορες ε, συναντήσεις παρέχοντες πολύτιμες πληροφορίες και ιδέες για τη σύνταξη του κειμένου. Λίγο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας. Άρα μια πανορομική άποψη θα σας δώσω του εγγράφου εργασίας. Είναι το δεύτερο έγγραφο. Εκπροσωπεί τα αποτελέσματα της φάσης των ερευνών, αλλά ε, αποτελεί επίσης την επεξηγηματική δήλωση της εκθέσεως αναφέρεται στα βασικά θέματα γύρω από τα οποία θα περιστραφεί το κείμενο. Αφετηρία δεν εκρύφτηκε από το προηγούμενο έγγραφο εργασία. Είναι πεποίθηση ότι η χάρτα αντιπροσωπεύει ακόμα σε πολλές περιστάσεις ένα ε, μεγάλο βασικό στοιχείο στη διαδικασία λήψη αποφάσεων Ευρωπαϊκής ενώσεω. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τους συνομιλητές με τους οποίους συζητήσαμε. Παρά τις διαδικασίες που έγιναν μετά από τη συνθήκη της Λισαβόνας, Υπάρχουν πολλές σκιώδες, σκιώδεις ζώνες και πολλά περιθώρια βελτιώσεων. Σε κάποιους τομείς η παιδεία δραστηριοτήτων είναι η ανάγκη πιο φανερή από τις άλλες. Και όπως είδαμε και στη φάση των ερευνών προσπαθήσα να επικεντρωθώ προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα που όμως θα αναφερθούν εκτενέστερα και λεπτομερέστερα στην έκθεση. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειε όσον αφορά τις διάφορες προτάσεις των διαφόρων το, για τους διάφορους τομείς. Ακροθυγός να σταθώ στα δύο σημαντικά όρια για την πλήρη λειτουργικότητα της χάρτας που από εκεί άμεσα δημιουργούνται τα εφαρμοστικά κενά. Πρώτα απ' όλα η συμπεριφορά των θεσμών έναντι της χάρτας. Τι διαφαίνεται. Μια παθητική ερμηνεία της χάρτας που έχει σαν στόχο τη μη παραβίαση των διατάξεων αυτής παρά την προώθηση της πλήρους υλοποίησης της χάρτας. Αυτό το είδαμε στις διάφορες φάσεις του νομοθετικού έργου και της ε, λήψης αποφάσεων της ενώσεως. Είναι μια συμπεριφορά που φαίνεται ότι δίνει στη χάρτα μία δευτερογενή νομιμοποίηση σε σχέση με τις συνθήκες. Όμως ε, βλέπουμε ότι απορρέει από, πρωτογενώς από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο η χάρτα. Υπάρχουν και όρια που απορρέονται από το άρθρο 51 της χάρτας. Από τη μία πλευρά έχουμε μια διχοτομία, όπως αποκαλείται, μεταξύ δικαιωμάτων που πρέπει να σέβεται κανείς και αρχών που πρέπει να τηρεί και απ' την άλλη το πεδίο εφαρμογής της χάρτας στα κράτη-μέλη. Και στις δύο περιπτώσεις η δραστηριότητα της έρευνας έδειξε τις δυσκολίες κατανόησης, πλήρους κατανόησης της λειτουργικότητας των διατάξεων. Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει αυτή η διχοτομία αρχών δικαιωμάτων και δημιουργεί και ερμηνευτικά εμπόδια όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων της χάρτας, αλλά δημιουργεί και κινδύνους σμίκρινσης της εμβέλειας της χάρτας. Και αυτό που διαφαίνεται από την ανάλυση της σχετικότητας των ηθικών αρχών που θα έπρεπε να είναι δικαιώματα στα πλαίσια της οικονομικής διακυβερνήσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Στη δεύτερη περίπτωση η πρακτική που ακολουθούν τα κράτη-μέλη καταδεικνύει σαφώς αμφίσιμη εφαρμογή των διατάξεων και αυτό οδηγεί σε μια χαμηλότερη, μικρότερη χρήση της χάρτας σε εθνικό επίπεδο που θα έπρεπε. Κλείνοντας, βλέπουμε, διαπιστώνεται ότι εμφανίζεται μια συνετή προσέγγιση της χάρτας, επιφυλακτική με περιοριστικές συνέπειες όσον αφορά την εφαρμογή και υλοποίηση των διατάξεων, ο επαναπροσδιορισμός, επαναπροσδιορισμός μάλλον των αρχών και μέσω α, νέου προβληματισμού επί του άρθρου 51, κατά την άποψή μου, είναι προαπαιτούμενο για να δοθεί πλήρης αξιοπρέπεια στη χάρτα και να αποτελεί απαρέγκλητη, απαρέγκλητη βάση για τα μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν ούτω ώστε να έχει πλήρη αποτελεσματικότητα η χάρτα αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Θα μιλήσει κανείς εκ μέρους του Έλμαρ. Δεν έχουμε τον Έλμαρ. Τη Σιλβί. Θα τα μιλήσετε. Η Σιλβί Κάουφμαν για του σοσιαλιστέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την Μπάρβαρα για την πολλή δουλειά που έχει κάνει στο σημαντικό αυτό θέμα. Νομίζω ότι τώρα με το έγγραφο εργασίας έχουμε ένα έγγραφο το οποίο μας δείχνει και την κατεύθυνση της μελλοντική έκθεσης. Ως σκιώδης εισηγήτρια θα ήθελα να ακούσω τα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση της έκθεσης, διότι δεν το γνωρίζω. Όσον αφορά το περιεχόμενο, Για παράδειγμα, τη... βρίσκω ότι η δουλειά με τον οργανισμό για τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα είναι πολύ σημαντική. Δεν νομίζω ότι εκμεταλλευόμαστε επαρκώς σε την ύπαρξη αυτού του οργανισμού. Επίσης, το θέμα του Ευρωπαϊκού Χάρτη Κοινωνικών Δικαιωμάτων είναι σημαντικό για να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών. το να έχουμε εμπειρογνώμονα για την εφαρμογή του χάρτη ε, κοινωνικών δικαιωμάτων και αυτό πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα. Ενός οργανισμού δηλαδή που θα ενεργεί ως εμπειρογνώμων. Επίσης, ε, λέει ότι οι μελέτες αντικτύπου ε, είναι άχρηστες στους τριμερείς διαλόγους. Εγώ δεν θα συμφωνήσω. Ήμουν εισηγήτρια για την βελτίωση της νομοθεσίας ε, και την διοργανική συνεργασία. Όταν δίδεται τόση μεγάλη σημασία στις μελέτες αντικτύπου και ουσιαστικά ε, υποδεικνύεται η κατεύθυνση στους πολιτικούς. Ε, αυτό δεν επιτρέπεται να γίνεται. Ε, οι μελέτες αντικτύπου είναι ένα απαραίτητο εργαλείο. Πρέπει να υποβάλλεται από, τις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν έχουμε προτάσεις νέας νομοθεσίας. Και εάν ε, θεωρήσουν τα θεσμικά όργανα ότι οι μελέτες αντικτύπου πηγαίνουν προς ε, τελείως αντίθετη κατεύθυνση, μπορούν να εκπονήσουν δικές τους. Μπάρμπαρα, σε ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά που έχεις κάνει. Ζητώ συγγνώμη, ε, διότι είχα ψηφοφορία και σε άλλη επιτροπή. Γι' αυτό πρέπει να φύγω, αλλά θα ήθελα πολύ να ακούσω τα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Προτού να δώσω το λόγο στον επόμενο ομιλητή, ε, θα ήθελα να σα ενημερώσω για το χρονοδιάγραμμα. Στι 21 Νοεμβρίου θα γίνει η παρουσίαση του ψηφίσματο μετά από την παρουσίαση του εγγράφου εργασία σήμερα. Κατόπιν έχουμε μια προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών πάνω στο σχέδιο ψηφίσματο 30 Νοεμβρίου. Τον Ιανουάριο θα εξετάσουμε τι τροπολογίε και τον Φεβρουάριο θα ψηφίσουμε στην ΑΦΚΟ. Το έγγραφο εργασία λοιπόν τη Μπάρμπαρα θα γίνει η αιτιολογική έκθεση έτσι λοιπόν θα το ψηφίσουμε και αυτό ουσιαστικά. Ε, Μάιτε, θες το λόγο. Κάποιος άλλος. Μόνο ευχαριστώ θέλω να πω. Ευχαριστώ πολύ. Δεν, βλέπω να ζητάει κανείς άλλος και όδηση ε, το λόγο. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να κλείσουμε το σημείο αυτό της ημερησίας διάταξης ε, και από ό,τι κατάλαβα η Μπαρμπάρα θα εκπονήσει τώρα το σχέδιο ψηφίσματος ε, μέχρι την επόμενη συνεδρίαση. Και συνάδελφοι, ε, στην προετοιμασία της έκθεσης αυτής είχαμε συνομιλίες με, το, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Νομίζω λοιπόν ότι η Μπάρμπαρα κάνει πολύ καλή δουλειά και θα συνεχίσει αυτό να είναι σημαντικό στοιχείο ε, στις συζητήσεις μας για το πώς η Ευρώπη μπορεί να εφαρμόσει καλύτερα ε, τον χάρτη θεμελιωτών δικαιωμάτων. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης, εφαρμογή των διατάξεων των συνθήκων σχετικά με την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάιτε, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το έγγραφο εργασίας παρουσιάστηκε στο Στρασβούργο την 1η Οκτωβρίου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να επαναλάβω όλα όσα είπαμε τότε. Όμως ευχαριστώ και τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι παρόντες για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή ασχολήθηκε με ζητήματα που έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτήν την έννοια που είναι η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και το 2017 και με το πρόγραμμα για τις αρχές και τις αξίες. Και τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι η Επιτροπή θέλει να ενισχύσει διάφορες δυνατότητες εφαρμογής της έννοιας αυτής της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Επίσης, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής τότε μας είχε πει ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να μπορούν και σε επόμενες ευρωεκλογέ κυρίως να ασκήσουν όλα τα δικαιώματά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες. Όπως λοιπόν λέμε και στο έγγραφο εργασία υπάρχουν περιορισμοί και αδυναμίες στην εφαρμογή ε, της ε, οδηγίας του 2004 για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Και πρέπει να πούμε πέρα δηλαδή από ό,τι άλλη δουλειά γίνεται για την εφαρμογή ό,τι συστάσει και αν κάνουμε στις διάφορες ανταλλαγέ απόψεων, διαπιστώνουμε πάντα ότι υπάρχει η σαφής ανησυχία από τον κόσμο σε σχέση με τι. Με την ερμηνεία, την αυστηρή ή όχι, της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Και σε σχέση μάλιστα και με την άνοδο του λαϊκισμού έτσι λοιπόν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σε ό,τι συζητήσεις είχαμε μέχρι τώρα, βλέπουμε ότι αυτό το θέμα έρχεται και επανέρχεται. Το πρόβλημα της διαπαιδαγώγησης του κόσμου για να ξέρει τι είναι η Ευρωπαϊκή Θαγένεια. Η καταπολέμηση των διακρίσεων Αντίθετα, ακούμε διάφορες συζητήσεις και πυρήνους λόγου που δεν έχουν καμία σχέση με το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει το ανήκειν σε μια πολιτική οικογένεια. Και μάλιστα στι συζητήσεις με τους συναδέρφους ακούμε ξανά και ξανά και βλέπουμε ότι υπάρχει ένα χάσμα μεγάλο ανάμεσα σε αυτό που πιστεύει ο κόσμο ότι είναι η Ευρωπαϊκή Θαγένεια και σε αυτό που πραγματικά είναι η Ευρωπαϊκή Θαγένεια και αυτό που μπορούμε εμείς να προσφέρουμε. Γιατί μερικές φορές εμείς ε, τα θέματα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας τα φύγουμε έτσι ακροθυγώς, ενώ ο κόσμος περιμένει από εμά έτσι πιο ορμητικά να μπαίνουμε σε αυτό το ζήτημα. Οπότε εγώ θα προσπαθήσω στην έκθεση αυτή να βάλω όσο περισσότερα πράγματα και να θέσω μπροστά στις ευθύνε τους όλους. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέρφους που συνεργάστηκαν μαζί μου. Τα βλέπουμε τα σημεία των καιρών. Η ευρωπαϊκή θαγένεια προσφέρει πολύ περισσότερες δυνατότητες και θα έπρεπε να τις χρησιμοποιήσουμε. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για όλα όσα σχολιάσατε που θα τα προσθέσω στο κείμενό μου. Ακριβώς επειδή οι πολιτικές συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε είναι αυτές που είναι, πρέπει να αποφεληθούμε στο έπακρον από αυτήν την ευρωπαϊκή θαγένεια και την έννοια της ευρωπαϊκής θαγένειας. Ελκ, Μπόνι και μετά η Μπάρμπαρα Σπινέλη. Δεν έχουμε άλλους σκιώδες, εντάξει. Και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Μαρία Ελέν Μπουλανζέρη είναι εδώ, σωστά. Λοιπόν, παρακαλώ. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το έγγραφο εργασίας. Δεν είχα τη δυνατότητα να συμμετάσχω σε προηγούμενες συζητήσεις. Συμφωνώ όμως απολύτως με πολλές από τις προτάσεις και συστάσεις της πρότασης αυτής. Νομίζω ότι είναι ένα ολοκληρωμένο και πλήρες έγγραφο εργασίας. όπου περιγράφεται σωστά το νομικό πλαίσιο που σχετίζεται με την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, τίθενται κάποια ερωτήματα σημαντικά για την περαιτέρω συζήτηση. Και νομίζω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό ότι τίθενται πολλά ερωτήματα στο έγγραφο εργασίας που θα μας βοηθήσουν να λύσουμε με πρακτικό τρόπο διάφορα προβλήματα, διότι δεν μιλάμε γενικά για την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλάμε για συγκεκριμένες δράσεις, για συγκεκριμένα προγράμματα που πρέπει να γίνουν για να δημιουργηθεί ένας καλύτερος χώρος, καλύτερα κίνητρα, καλύτερες συνθήκες για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ιθαγένειας Και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι θα πρέπει να αποφύγουμε και κάποιες συγκεκριμένες πιέσεις. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για την εκπαίδευση. Το πώς θα εκπαιδευτεί κανείς να είναι Ευρωπαίος πολίτης. Ε, κάποιοι λένε ότι αυτά είναι αρμοδιότητες ε, των κρατών μελών. Νομίζω όμως ότι είναι απαραίτητο ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση να ενσωματώσουμε στην εκπαίδευσή μας εκπαίδευση και για την ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Τι σημαίνει, πώς λειτουργεί, τι πλειονεκτήματα έχει κανείς από αυτήν, διότι νομίζω ότι αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεύτερο θέμα είναι το πώς μπορεί να ασκεί κανείς τα δημοκρατικά του δικαιώματα. Αυτά είναι, αυτό είναι ένα από τα θέματα κλειδί για την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την άσκηση των δημοκρατικών μας δικαιωμάτων. Είναι σημαντικό αυτό να γίνεται αφενός ε, στα κράτη-μέλη μας απέναντι στους ε, θεσμούς εκεί, ε, αλλά και απ' την άλλη πρέπει να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πώς λοιπόν να ενθαρρύνουμε την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την συμμετοχή, διότι η λέξη κλειδί για τους συνειδητοποιημένους πολίτες είναι ακριβώς η συμμετοχή. Στην έκθεση περιλαμβάνονται κάποιες προτάσεις για το τι προγράμματα μπορούμε να εφαρμόσουμε, πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις σύγχρονες τεχνολογίες, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Και τώρα που συζητάμε υπό το φως του μελλοντικού πολιετούς δημοσιονομικού πλαίσιου, ε, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα προστιθέμενης αξίας, διότι είναι σημαντικό στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα στο τοπικό επίπεδο, να δώσουμε λοιπόν σε αυτούς κάποια εργαλεία, κάποιους οικονομικούς πόρους για να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για άσκηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και δημιουργίας αυτού του δημοσίου χώρου ώστε να μπορέσουμε να ενώσουμε, να συνδυάσουμε την εθνική μας ηθαγένεια με την ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσβλέπω λοιπόν την καλή συνεργασία με την Μάιτε και τους άλλους σκιώδεις εισηγητές πάνω στο έγγραφο αυτό. Δεν θα περιγράψουμε μόνο το νομικό πλαίσιο, Δεν θα περιγράψουμε μόνο το νομικό πλαίσιο και κάποιες συγκεκριμένε ε, δράσεις και προγράμματα, αλλά θα αναφέρουμε ότι η Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα από τα θέματα κλειδί για την προάσπιση της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Και εάν κάποιοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει ε, δημοκρατία, να αναπτύξουμε την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Μπάρμπαρα, παρακαλώ. Θα ήθελα να, να σε ευχαριστήσω για τις συστάσεις που έκανες. Υπάρχει ένα σημείο που πολύ με ενδιαφέρει. Αυτό αφορά τους εθνικισμούς. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι είναι μια πρόσκληση, μια έκκληση να μην περιοριστούμε στο να καταγγέλουμε το φαινόμενο και να πούμε δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες της ενώσεως, αλλά να πάμε στο στις να καταλάβουμε τις ρίζες του πολλαπλασιασμού, του εθνικισμού. Να καταλάβουμε σε ποιο βαθμό αυτό το φαινόμενο αποκαλύπτει ευθύνη των δυνάμων, των δυνάμων που μέχρι τώρα κατεύθυναν την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι μας μαθαίνει η ιστορία ότι αν αυτά τα φαινόμενα της δημοκρατίας δεν αναλυθούν αλλά απλώς καταγγελθούν και καταδικαστούν στο τέλος έχουμε σοβαρότερες κρίσεις. Η ιστορία της δημοκρατίας της Βαϊμάρης το αποδεικνύει σαφέστατα. Το κλειδί κατά την άποψή μου είναι στην έκφραση που χρησιμοποίησε η Μαϊτέ της προωθημένης ενισχυμένης ηθαγένειας, της προβεβλημένης ηθαγένειας. Κατέληξα στο συμπέρασμα από τις εργασίες ε, της χάρτας. Τα δικαιώματα όπως και η ηθαγένεια είναι στοιχεία που θα πρέπει να τα υπερασπιστούμε και να τα προωθήσουμε. Α, στα άλλα σημεία που ανέφερε η συνάδελφος Μπόνη, τα σημεία αυτά που ανέφερε είναι σημαντικά για μένα και η ιδέα της ε, συμμετοχής στα πολιτικά δρόμενα, στην, συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών χρειάζεται για να αντιμετωπιστεί μια δημοκρατική κρίση. Μια, μια, μια κρίση των συνδικάτων, των κομμάτων, όλων των ενδιάμεσων φορέων της κοινωνίας και αυτή η αδυναμία των ενδιαμέσων αυτών φορέων δημιουργεί αυτά τα φαινόμενα του εθνικισμού, κρίση των ευρωπαϊκών θεσμών που βλέπουμε, που διαπιστώνουμε σε όλη την Ένωση. Ευχαριστώ και ευχαριστώ Μαϊτέ θα συνεργαστώ στο βαθμό των δυνατοτήτων μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Γιώ Λάινεν για τους συντονιστές που αντικαθιστά τον Πέντρο Σίλβα Πρέντα. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. θα σας διαβάσω τις παρατηρήσεις ε, του Αντιπροέδρου μας ε, του κυρίου Περέιρα φυσικά θέλει να συνεργαστεί μαζί σας, ε, στηρίζει την βασική κατεύθυνση του εγγράφου εργασίας. Λέει τα εξής. Τα ευρωπαϊκά μέσα στη διάθεσή μας υπό το παρόν πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο δείχνουν ότι οι ε, Ευρωπαίοι πολίτες, ιδιαίτερα οι νέοι Ευρωπαίοι, ενδιαφέρονται για το θέμα της ηθαγένειας. Και γι' αυτό το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να ε, λάβει υπόψη αυτό το γεγονός, χρηματοδοτώντας νέα προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη και την ε, ανάγκη ε, να ασχοληθούμε με τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, θα πρέπει το θέμα της ηθαγένειας να είναι ο πυρήνας όλων των νομοθετικών μας εργασιών. Και αυτό συνάδει με τις πιο πρόσφατες νομοθετικές μας ενέργειες. Πέρα από το να εξετάσουμε την κατάσταση όσον αφορά την ευρωπαϊκή ηθαγένεια, θα πρέπει να ευθυγραμμιστούμε με κάποιες σημαντικέ ε, εκθέσεις πρωτοβουλία που συζητώνται αυτή τη στιγμή στην ε, ΑΦΚΟ, όπως είναι η έκθεση ΑΟΡΕΚΙ για το ε, μέλλον της Ευρώπης, την δική μου έκθεση για την διαφάνεια στο Συμβούλιο και την έκθεση για την καλύτερη νομοθεσία. Μεταξύ των προτεραιοτήτων που μπορούμε να αναφέρουμε μέχρι το τέλος της θητείας αυτής, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικός ο στόχος ε, ενθάρρυνσης της συμμετοχής των πολιτών στις ευρωεκλογές. Επίσης, είναι υψίστης σημασίας να δράξουμε την ευκαιρία να ζητήσουμε μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ενίσχυσης της συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών στις ευρωεκλογές. Εκτιμούμε την σημαντική αναφορά στο έγγραφο εργασίας της εκπαίδευσης. Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε έναν ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο και να δείξουμε τις πραγματικές διαστάσεις της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Αυτό ε, συνδυάζεται με την ανάγκη εις βάθος εργασίας σχετικά με την ανάγκη της παιδαγωγικής και της εκπαίδευσης σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών. Επίσης, υπάρχουν 50 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών που ζουν σε άλλο κράτος μέλος ε, από το δικό τους και για αυτούς χρειάζονται δράσεις για να ξεπεραστούν οι διάφορες μορφές διακρίσεων ε, που ε, υπάρχουν. Θα ήταν χρήσιμο να ξεκινήσουμε συζήτηση με μη κυβερνητικέ οργανώσει για να δημιουργήσουμε έναν ευρωπαϊκό φορέα που να εκπροσωπεί τους ε, πολίτες αυτούς και να υπερασπίζεται τα δικαιώματά τους. Και κλείνοντας, άλλο ένα θέμα είναι και ο σεβασμός της πολυγλωσσίας υπάρχουν ακόμη εμπόδια τα οποία πρέπει να ξεπεράσουμε όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες επιγραμμικά και στον πραγματικό κόσμο. Αυτές λοιπόν ήταν οι παρατηρήσεις του Σίλβα Περέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ο ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεισέφεραν σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον έγγραφο. Κατά παράδοση, η ηθαγένεια έχει να κάνει με τη φορολογία. Και ε, ε, με τη στρατιωτική θητεία. Αλλά αυτό έχει αλλάξει τώρα στον 21ο αιώνα. Τώρα ε, έχει να κάνει με την πολύπλοκη σχέση ανάμεσα στην κρατική εξουσία και τους πολίτες. Αυτό φυσικά σχετίζεται με προβλήματα λογοδοσίας, ε, το θέμα της συγκατάθεσης για την άσκηση της εξουσίας ε, και ε, την εξουσιοδότηση. Και εδώ έχουμε τις δυσκολίες. Πώς μπορεί λοιπόν εδώ να δημιουργήσει κανείς θεσμικά όργανα που να δείχνουν στους πολίτες ότι μπορούν να επηρεάσουν αυτά που κάνουν τα θεσμικά όργανα. την αίσθηση δηλαδή ότι εξουσιοδοτούνται από τους πολίτες ε, τα θεσμικά όργανα και η κοινωνία των πολιτών μπορεί ε, να χειροτερεύει τα πράγματα διότι αποκλείει κάποιους πολίτες. Η κοινωνία των πολιτών δεν μπορεί να εκπροσωπεί όλους τους πολίτες, μόνο κάποια επιλεγμένα τμήματα ε, του πληθυσμού μπορεί να εκπροσωπεί. Πώς λοιπόν μπορούμε να δημιουργήσουμε φορείς για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Αυτό νομίζω είναι κεντρικής σημασίας εάν θέλουμε να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Ερώτηση. Τι υποχρεώσεις συνοδεύουν την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Η ιθαγένεια αυτή, ε, αν σχετίζεται μόνο με δικαιώματα και όχι με υποχρεώσεις, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει τελικά. Και τέλος, το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται στους νέους. Ωραία και καλά, όλοι είμαστε υπέρ αυτού, αλλά να έχετε κατά νου ότι ε, η μεγαλύτερη κατηγορία πληθυσμού μάλλον ε, σύντομα θα βρίσκεται άνω των 65 ετών. Θα πρέπει λοιπόν ε, να εξετάσουμε και το θέμα της άσκησης των δικαιωμάτων των πολιτών άνω των 65 ετών. Εάν το 50 ή 60% του πληθυσμού ε, είναι άνω της ηλικίας των 65, θα έχει τελείως διαφορετική μορφή η κοινωνία. Και αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία κινείται η Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλέσαμε να συμμετάσχετε σε ένα διάλογο. Ε, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμμετάσχουν μαζί μας. Η κυρία Μαρία Ελέν Μπελανζέ, που είναι τμήματάρχη τη Γενική Διευθύνσεω για θέματα δικαιοσύνη, ασχολείται πιο συγκεκριμένα με την ηθαγένεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει κάποιος, είστε εκεί. Έχετε το λόγο. Μπορείτε να παρουσιάσετε εν συντομία τις ε, πολιτικές που εφάρμοσε η Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Αλλά αν θέλετε και να σχολιάσετε είσαστε ευπρόσδεκτοι. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, για τις σημαντικές συνομιλίες. Η ηθαγένεια είναι στην καρδιά των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ενώσης, αναφέρθηκε. Στις συνθήκες αναφέρεται και παγιώνεται. Η ελεύθερη διακίνηση είναι ένα από τα βασικά δικαιώματα που θεσπίζει. Η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές, τοπικές εκλογές, δικαίωμα ε, προστασίας προξενικής, συμμετοχή στο Ευρωκοινοβούλιο, να προσφεύγει κανείς στο συνήγορο του πολίτη. Ε, είναι πολύ σημαντικό δικαίωμα ευρωπαϊκό που πηγαίνει με την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Θα θυμόσαστε ότι το 2015 αυτή η Επιτροπή μαζί με άλλες τρεις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διοργάνωσαν μια ακρόαση όσον αφορά την ευρωπαϊκή ηθαγένεια σημαντικότατο βήμα για να ετοιμάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έκθεση περί ηθαγενείας. Βάσει το άρθρο 25 των συνθήκων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε τρεις-τρία χρόνια υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για την πρόοδο που επετεύχθη όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Και το άρθρο 25 της συνθήκης ε, προβλέπει ενίσχυση των δικαιωμάτων μέσω συγκεκριμένη διαδικασίας να έχει πρόσβαση στα δικαιώματα αυτά. Είναι συγκεκριμένες διαδικασίες, δεν είναι αλλαγή των συνθήκων. Η πρόσφατη έκθεση που εξέδωσε για την Ιθαγένεια Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξεδόθη μετά την ακρόση. Η έκθεση γίνει το 2017 ήταν αυτή αναφέρει ότι ασκούν όλο και περισσότερο οι πολίτες τα δικαιώματα της Ιθαγένειας Ευρωπαϊκής όπως είπατε στην παρέμβαση, στον αριθμό των κινουμένων πολιτών, των μετακινουμένων πολιτών τη ευρωπαϊκή ενώσή. Όλο και περισσότεροι γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους, στο καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Πρέπει ε, ε, να γνωρίζουν καλύτερα οι πολίτες τα δικαιώματα και να εφαρμόζονται τα δικαιώματα. έκθεση βασίστηκε στις διάφορες πηγές, το είπαμε και στην ακρόαση και είχαμε και τροφοδότηση άμεσα από τους πολίτες. Ε, παρενέβησαν πολλοί οι πολίτες, εξέφρασαν απόψει για την ηθαγένεια, πηγαίνουν, προσφεύγουν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το ευρωβαρόμετρο το δείχνει αυτό και άλλες στατιστικές. Να αναφέρω ακροθυγώς κάτι. Κάποιες από τις δράσεις που ακολουθούμε για να προωθήσουμε ε, αυτά τα δικαιώματα. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τα δικαιώματα τη ηθαγένεια παρουσιάσαμε φέτος πρόταση για ε, τέτοια ταυτότητας για τους μετακινούμενους και διάφορα ταξιδιτικά έγγραφα που βοηθούν στην ε, μετακίνηση των πολιτών. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των εγγράφων και το πώ γίνονται αποδεκτά από άλλα κράτη-μέλη αυτά τα ταξιδιτικά εγγράφα. Αυτό είναι κάτι που το εξετάζει αυτό το Κοινοβούλιο και συζητείται και στο Συμβούλιο. Είναι θέμα συναπόφαση. Επίσης ε, παρουσιάσαμε φέτος ε, μια έκθεση για την άσκηση των δικαιωμάτων ε, ψηφο, ψήφου σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά και υπάρχουν πολλές καλές πρακτικές που υπόσχονται πολλά. Τις επεξεργαζόμαστε τις καλές πρακτικές, ήδη αναφέρθηκε. χρειάζεται θέμα να, προωθήσουμε το πρόγραμμα για την ισότητα και βοηθάμε τους φορείς που προωθούν την άσκηση των δικαιωμάτων. Και υπάρχει και πρόγραμμα ενδιαφέρον. Συμμετέχουν διάφορες πόλεις. Ανταλλαγή των πρακτικών κάνουν για το πώς κινούνται στο κατάλληλο δίκτυο. Κάθε χρόνο διοργανώνουμε εργαστήριο. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ιθαγένειας, αυτή είναι η εβδομάδα, θα συζητήσουμε σε τοπικό επίπεδο την άσκηση των δικαιωμάτων, κυρίως των εκλογικών δικαιωμάτων και τη συμμετοχικότητα σε τοπικό επίπεδο. Θα ξέρετε όλοι ότι φέτος είχαμε πολύ σημαντικό γεγονός για την Ιθαγένεια, νέα οδηγία για την προστασία καταναλωτών. Και αυτό είναι κομμάτι των δικαιωμάτων που απορρέουν την Ιθαγένεια. Αυτή η οδηγία ετέθησε ισχύ φέτος. Παρακολουθούμε την εφαρμογή, την υλοποίησή της και παρακολουθούμε προσεκτικά τι γίνεται στα κράτη-μέλη όσον αφορά την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας. Και διάφορες δραστηριότητε κάναμε για να προωθήσουμε τα δικαιώματα. Φέτος, εκστατεία ενημέρωση διοργανώσαμε για το δικαίωμα προστασίας καταναλωτού, το δικαίωμα που έχει κανείς όταν χρειαστείς να πας άλλο κάτω μέλος και δεν έχεις κάποιο ε, εκπρόσωπο της χώρα σου εκεί και κατεπήγον έγγραφο ανάγκη, ταξιδιωτικό έγγραφο, αν χάσει το ταξιδιωτικό σου έγγραφο στο εξωτερικό, μπορεί να πα σε προξενική αρχή και να πάρει κάποιο έγγραφο. Έχει, υπάρχει πρότυπο έντυπο και προτείναμε να εξυγχρονιστεί για να διευκολυνθούν οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα του αν έχουν χάσει τα έγγραφά του. Έχουμε και ρήτρα προξενική προστασία. Οι Ευρωπαίοι πολίτε να μπορούν να ωφεληθούν από το δικαίωμα προξενική προστασία Τέλος, εξίσου σημαντικό, χωρίς να μακρηγορήσω, να πω κάποια πράγματα τώρα για τα εκλογικά δικαιώματα. Σημαντικότατη είναι η εξέλιξη σε αυτό το πλαίσιο. Το ξέρετε πολύ καλά. Είναι πρόταση του Κοινοβουλίου. Ο εκλογικό νόμο Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκή Ενώση μεταρρυθμιστεί από την πλευρά μα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, εξασφαλίζουμε ότι δίδονται σωστέ πληροφορίε για την άσκηση των δικαιωμάτων. Ίσως είναι πολύ τεχνικό το θέμα, αλλά είναι σημαντικό να ενημερώνεται σωστά ο κόσμος. Πώς μπορεί να ε, εγγραφεί, να ασκήσει τα εκλογικά του δικαιώματα. Συνεργαζόμαστε γι' αυτό με τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να κυκλοφορούν σωστές πληροφορίες. Προτείναμε φέτος πολλές ε, πρωτοβουλίες για να προθήσουμε τη σωστή συμπεριφορά, τη σωστή διεξαγωγή των ευρωεκλογών Είχαμε πρόσφατη πρόταση που κάναμε. Πακέτο προτείναμε. Ελεύθερες και δίκαιε εκλογές, διεξαγωγή ελευθέρων και δικαίων εκλογών. Παρουσίασε το πακέτο τον περασμένο μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμπεριέχονται διάφορα στοιχεία στη δέσμη μέτρων. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι κανεί δεν μπορεί να ωφεληθεί από παραβίαση παραβιάσεως δεδομένων για να επηρεάσει τη διεξαγωγή των εκλογών. Υπάρχει κάποια σύσταση Βάσει αυτή πρέπει να συνεργαστούν τα κράτη-μέλη εσωτερικά, οι διάφορες αρχές και τα κράτη-μέλη μεταξύ τους να συνεργαστούν για να προστατεύσουν την κεραιότητα των εκλογών και σύσταση προς τα κράτη-μέλη και τα πολιτικά κόμματα απευθύνεται για την αύξηση της διαφάνειας ούτω ώστε όταν ψηφίζει ο κόσμος να γνωρίζει ποιο επικοινωνεί μαζί τους ότι αυτό το πολιτικό μήνυμα που τους στέλνουν, από πού προέρχεται, από πού χρηματοδοτείται το κόμμα. Επίσης να υπάρχει προστασία από κυβερνοεπιθέσεις και κυβερνοαπειλές και να γίνουν κάποιες δραστηριότητε ευαισθητοποίησης από τα κράτη-μέλη. Είναι πολύ σημαντικό πακέτο. Ένας από τους σκοπούς του πακέτου είναι να καταπολεμηθεί η παραπληροφόρηση στα πλαίσια των επικειμένων ευρωεκλογών. Δεν θα είμαι εξαντλητική, υποσχέθηκα ότι δεν θα μακρηγορήσω. Να πω Έχουμε ένα συμπόσιο προετοιμάσει, πολύ σημαντικό, τέλος Νοεμβρίου. Συμπόσιο υψηλού επίπεδου περί δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε πολλά από τα σημεία που αναφέρθηκαν σήμερα. Με τα χαράς να απαντήσω. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι θα συνεχίσουμε το διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Γραμματεία ετοιμάζει μια τεχνική ε, φύσεως συνάντηση με την κυρία Μπουλανζέρ για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε εκτενέστερα απόψει για αυτά τα στήματα και εννοείται ότι θα καλέσουμε την εισηγήτρια του Σκιώδης αλλά και τους συντάκτες γνωμοδότησης από τις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές και όσοι συνάδελφοι θέλουν να συμμετάσχουν Ευχαριστώ. Μάιτε, σύντομα αν μπορείτε για να κλείσει το θέμα αν χρειάζεται. Αλλά, α, η Μπάρμπαρη ήθελε να πει κάτι. Σύντομο όμως, ε. Πάρα πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα. Να πω κάτι πάνω σε αυτά που είπε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σημαντικό σημείο. Η προστασία η προξενική για τους πολίτες. Ευπρόσδεκτες οι οδηγίες, οι καινούριε ή οι πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στα διάφορα κράτη-μέλη. Ξέρω ότι η προξενική προστασία στην περίπτωση της Ιταλίας έχει εξαφανιστεί ουσιαστικά. Οι βασικές υπηρεσίες όπως ε, διάφορα έγγραφα πρέπει να εκδίδονται ε, ε, ανατίθενται υπό υπεργολαβία, επιπληρωμή και αυτό λόγω περικοπών του προπολογισμού. Αυτό είναι σημαντικό όσον αφορά την προξενική προστασία για τους ε, πολίτες. Ναι, πολύ ενδιαφέρον και αυτό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάιτε τώρα, σε ένα λεπτό αν μπορείς. Ευχαριστώ. Ε, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας όλους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά λοιπόν την προξενική προστασία συγκεκριμένα, στην Ειδική Επιτροπή για την Τρομοκρατία δουλεύουμε για την εκπόνηση συμφωνιών στα προξενία, γιατί όταν γίνει μια τρομοκρατική επίθεση σε μια χώρα μέλος και υπάρχουν εκεί πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμένη χώρα, υπάρχουν ένα σωρό προβλήματα. Είτε επιζήσει είτε όχι ένα άτομο από μια τρομοκρατική επίθεση και δεν βρίσκεται στη χώρα του, τα προβλήματα, είτε πρόκειται για την ψυχολογική υποστήριξη, είτε πρόκειται για τη μεταφορά, είτε πρόκειται για την επικοινωνία με τους συγγενείς. Είναι ζητήματα πάρα πολύ σημαντικά. Και αν είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαβαίνετε ότι τα προβλήματα ε, αυξάνονται εκθετικά. Γι' αυτό λοιπόν ήθελα να σας το πω να ξέρετε ότι είναι πράγματα τα οποία απασχολούν την Ειδική Επιτροπή για την Τρομοκρατία, να το ξέρετε. Τώρα ένα γενικότερο σχόλιο. Εδώ συζητάμε για την στήριξη του δημοκρατικού συστήματος απέναντι σε νέους κινδύνους και νέες απειλές. Είναι μια πολύ σημαντική έννοια έτσι που βρίσκονται στην καρδιά των πάντων, παρόλα αυτά βρίσκεται σε αδυναμία. Άρα μένει πολύ δουλειά ακόμα να κάνουμε. Ο δρόμος είναι μακρύς. Ευχαριστούμε κυρία Μπουλανζέ. Θέλετε να αντιδράσετε ή το σημειώνετε. Εντάξει. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και να σας ε, πω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι λίγη η θητεία μας όπου να είναι. Προτείνουμε 21 Νοεμβρίου το σχέδιο έκθεσης, 29 προθεσμία για υποβολή τροπολογιών, 6 Δεκεμβρίου εξέταση των τροπολογιών και έγκριση Ιανουάριο ή Φεβρουάριο στην Επιτροπή μας και στη ΛΥΜΠΕ. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα θα συνοηθούμε με τη Γραμματεία και την ΜΑΙΤΕ να δούμε αν πρέπει να υπάρξει κάποια αλλαγή. Και περνάμε γρήγορα στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι κάτι που έχει ετοιμάσει η Mercedes Μπρέζο. Πρόκειται για την έκθεσή της όσον αφορά τον ε, κοινοβουλευτικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τη Λισαβόνα, διδάγματα και τα επόμενα βήματα. Εδώ έχουμε καλέσει εμπειρογνώμονες να μας παρουσιάσουν τις απόψεις τους για την κατάσταση πραγμάτων και για το πώς ε, εκτελείται αυτός ο κοινοβουλευτικός έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Κομισιόν. Έχουμε το Διευθυντή του Τμήματος Πολιτικών και Διοικητικών Σπουδών τον, και καθηγητή στο Κολέγιο της Ευρώπης στην Ολυβία Κώστα και την ε, κυρία Εύα Μαρία Πόρτσεβα, η οποία το μόνο που έχω εδώ είναι ότι είσαστε διδάκτος στο δαγματικό δίκαιο, αλλά φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και άλλα να προσθέσετε, μπορείτε να μας τα πείτε. Και μετά από τους δύο πυρογνώμονες θα έχουμε και την παρουσίαση μελέτης από τον Μίλαν Ρέμακ μελέτη σχετικά με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ερευνητική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χρόνο όμω δεν έχουμε πολύ, όπως ξέρετε, οπότε σας παρακαλώ να είσαστε σύντομοι. Θα αρχίσουμε τους δύο πυρογνώμονες. Δεν ξέρω ποιος θέλει πρώτα να πάρει το λόγο. Ο κύριος Κώστα. Α, η Μερσέντε πρώτα, βέβαια. βέβαια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευπρόσδεκτοι φιλοξενούμενοι μας, ε, ευχαριστούμε που δέχτηκαν την πρόσκλησή μας. Θα έχω την ευκαιρία αργότερα να παρουσιάσω τις εργασίες μας. Θα ήθελα να επενθυμίσω στους συναδέλφους ότι στην έκθεση αυτή προβλέψαμε αυτή την πρώτη ακρόαση με δύο φιλοξενούμενους που θα αναφερθούν στα διάφορε πτυχέ του πολιτικού ελέγχου από πλευρά του Κοινοβουλίου επί τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Και αναθέσαμε και μία μελέτη που εξετάζει νομικά ποια είναι η κατάσταση. Τι μας ενδιαφέρει ουσιαστικά. Όχι μόνο δούμε ποια είναι τα διαθέσιμα μέσα, αλλά να λάβουμε υπόψη και τις εξελίξεις, τις συγκεκριμένες, όσον αφορά τη χρήση των ελόγω μέσων. Να δούμε πώς χρησιμοποιήθηκαν, υπό ποιες συνθήκες, ποια χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο από άλλα. Και γι' αυτό καλέσαμε την κυρία Πότσεβα να μας μιλήσει για το άλλο θέμα. Μία πτυχή είναι ο έλεγχος με σκοπό κυρώσεις, τιμωρητικός έλεγχος αν το πούμε έτσι, νομικός όρο που είναι κάπως υπερβολικός. Ε, είναι προτάσει μομφή, Φερρυπίν, η απόσυρση ψήφου εμπιστοσύνη, το δικαίωμα διεξαγωγή έρευνα, ο έλεγχος των κατεξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων, προφορικές ερωτήσεις, γραπτές ερωτήσει ούτω καθεξής. Ένα θέμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι η εξέλιξη του πολιτικού έλεγχου επί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό μέσω της διευθύνουσας εποπτείας, steering oversight, διαφορετικού είδους ελέγχου που εφαρμόζεται μέσω πρωτοβουλειών, που είναι αντικείμενο συνένεσης. Είναι πιο συνενετικός έλεγχος ξεκινά από την εποπτεία της διαδικασίας του προϋπολογισμού, έλεγχο της υλοποίησης της εφαρμογής νομοθεσίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιέχεται μια ενδιαφέρουσα πτυχή, διότι έλεγχος επί κλάδου από πλευράς ε, Ευρωκοινοβουλίου δεν επιτρέπει πλήρη έλεγχο επί της εκτελέσεως των πράξεων, των διατάξεων. Ένα τμήμα της εκτέλεσης ανατίθεται του εκτελεστικού έργου, ανατίθεται στις εθνικές κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια για νομοθεσία και σε κάποιες περιπτώσεις ε, στα κοινοβούλια, τα περιφερειακά και την τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα στοιχείο ε, είναι αυτό που δημιουργεί περιπλοκότητα όσον αφορά την εποπτεία της εκτέλεσης. Και από αυτού ζητήσαμε από την κυρία Πότσεβα που έχει επεξεργαστεί συγκεκριμένα το θέμα, να έρθει και να μιλήσει γι' αυτό. Ιδού λοιπόν είναι δύο διαφορετικέ πτυχές και υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα που θα αποτελέσει αντικείμενο ενός τμήματος της έκθεσης και συνδέεται με διάφορες εργασίες που κάναμε όσον αφορά τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια και τα περιφερειακά κοινοβούλια και το απόγευμα θα έχουμε μια τέτοια συνάντηση που δείχνει πόσο αυτή η πτυχή του ελέγχου της εκτελέσεως της νομοθεσίας είναι σημαντικό. Δηλαδή να εξετάσουμε και ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Κοινοβουλίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Λίγο πολύ αυτά είναι τα σημεία που περιμένουμε να αναφέρουν οι φιλοξενούμενοι μας και του ευχαριστώ για άλλη μια φορά που δέχτηκαν την πρόσκλησή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Κώστα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τη Mercedes Μπρέσο που μας κάλεσε. Θα μιλήσω γαλλικά και θα προσπαθήσω να μην μιλάω πολύ γρήγορα για να διευκολύνω τους διερμηνείς λιομιλητής. Μιλάμε για τον έλεγχο, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εγώ θα το δω πιο συνολικά, μια που έχουμε την εξαίρετη έκθεση του EPRS, που μπαίνει στις λεπτομέρειες. Εγώ γενικότερα θα μιλήσω για τη λογική του ελέγχου που είναι θεμελιώδης βέβαια στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αποτελεί ουσιαστικά και το λόγο υπαρξής του. Τι είδου έλεγχο τώρα και πρέπει να αναρωτηθούμε τι σχέσεις υπάρχουν ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ποιες είναι οι δυνατότητες που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ασκήσει αποτελεσματικό έλεγχο και πόσο αποτελεσματικός είναι αυτός τελικά. Αυτή είναι μια μεγάλη βέβαια προβληματική. Αναφέρθηκε και η εξότιμη βουλευτή πριν πώς γίνεται ο έλεγχος αυτός, ζητάμε λογαριασμούς, γίνονται συζητήσει, κυρώσεις κτλ. Έχει να κάνει και με το πολιτικό καθεστώς της Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αναρωτηθούμε και τι θεσμικό μπρικολάζ γίνεται εδώ και 30 χρόνια με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπορεί να αυξήσει την ε, δυνατότητα κοινοβουλευτικού ελέγχου που έχει. Εννοείται ότι ο έλεγχος δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο για όλα τα πράγματα, γιατί εξαρτάται και από τις θεσμικές σχέσεις. Αν δούμε λοιπόν λιγάκι τον έλεγχο, γενικά μιλώντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούμε να πούμε ότι καταρχήν ήταν πολύ ο έλεγχος αυτός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν μια υπηρεσία ε, που ε, προσλάμβανε εμπειρογνώμονες, που ορίζονταν και δεν λογοδοτούσαν στις ε, αρχές, αλλά που ήταν υποχρεωμένη να θέτει σε εφαρμογή τις ε, αρχές και τις αποφάσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν παρενέβαινε καθόλου στον ορισμό των μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ήταν περισσότερο η δράση του, πώς το πω, κυρωτική ποινική, όπως γίνεται συνήθως με τις γενικές συνελεύσεις και αυτούς που λογοδοτούν σε αυτές. Η ευθύνη έτσι καλώ συζητιόταν μια φορά το χρόνο όταν η αρχή παρουσίασε τις δραστηριότητές της στην κοινοβουλευτική συνέλευση. Γι' αυτό λέω ότι συνδέεται λιγάκι με τον επιχειρηματικό κόσμο και όχι με την κοινοβουλευτική πρακτική. Αυτά στην αρχή. Τώρα στη συνέχεια σιγά σιγά άρχισε να εμπλέκεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και περισσότερο στον ορισμό των ε, μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρχισε να ενισχύεται και ο έλεγχος και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσπαθώντας να μιμηθεί τα εθνικά κοινοβούλια, αποκτάει όλα τα ελεγκτικά εργαλεία που αναφέρονται και λεπτομερώς στην έκθεση που έχει υποβληθεί του EPRS. Βλέπουμε ότι στην πράξη στην πρακτική μάλλον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν δύσκολο να διακρίνουμε τις ελεγκτικές δραστηριότητες από τις άλλες, τις νομοθετικές, τις δημοσιονομικές. Όλες αυτές οι δραστηριότητες συμπληρώνονται, αλληλοσυμπληρώνονται, γιατί ο έλεγχος γίνεται και όταν εγκρίνεται ο προπολογισμό και όταν επαληθεύεται η εκτέλεση του προπολογισμού, η χρήση του και όταν ασχολούμαστε με την επιτροπολογία, τις εκτελεστικές πράξεις ή συζητάμε τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό και η έκθεση του PRS εξετάσει το θέμα ευρέως. Η άλλη αλλαγή ήταν η συνθήκη του Μάστριχτ και της Λισαβόνας, όπου ενισχύθηκε ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιλογή του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ε, Επιτρόπων. Με αποκορύφωμα τους Σπίτσε Κατιντάτεν τους επικρατέστερους υποψήφιους για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σήμερα ακόμα όμως μπορούμε να δούμε δύο τελείως διαφορετικά, με δύο διαφορετικούς τρόπους τη συνθήκη. Πρώτα υπάρχει λογική της υπηρεσίας, του οργανισμού. Έτσι βλέπουμε, μπορούμε να δούμε μάλλον την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν πρέπει να έχει εντελώς ελεύθερα τα χέρια να κάνει ό,τι θέλει και να μπορούν να υπάρχουν και κυρώσεις που υπάρχει η διαδικασία μομφής που προβλέπεται. Υπάρχει όμως και η λογική ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που λαμβάνει υπόψη περισσότερο την κυβερνητική φύση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία αρχίζει και θυμίζει όλο και περισσότερο μια κυβέρνηση και όλο και λιγότερο έναν οργανισμό, μια υπηρεσία. Είναι λοιπόν δύο λογικές που βέβαια εγγράφονται μέσα στη δημοκρατική διαδικασία που πρέπει να τηρείται η διάκριση των εξουσιών και είναι αλήθεια ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαλύεται, αλλά ασκεί αυστηρό έλεγχο επί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιορισμένο όμως. Οπότε η μομφή δεν αποτελεί πολιτικό μέσο, είναι ένα μέσο ποινικό, όπως το impeachment στις Ηνωμένε Πολιτείε και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καθαίρεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δεύτερη λογική είναι η κοινοβουλευτική, στην οποία γράφεται περισσότερο η ιστορία αυτή των Spitzenkandidaten και όπου το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή συνδέονται μέσω μιας πολιτικής λογικής, συνεταιριστικής και αυτό φάνηκε περισσότερο μετά τις εκλογές του 2014. Και σε αυτή τη δεύτερη λογική διαπιστώνουμε ότι ασκεί πολιτική το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάνω σε αυτά τα οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με έναν ε, μηχανισμό ο οποίος ε, μπορεί να οδηγήσει στην άρση της εμπιστοσύνης του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή. Σε όλες τις κοινοβουλευτικές σύγχρονες δημοκρατίες πάντως είναι η πλειοψηφία που τα λέει όλα αυτά. Δεν είναι το κοινοβούλιο που ελέγχει την κυβέρνηση, είναι κατά κάποιο τρόπο η κυβέρνηση που υπερισχύει, ακριβώς επειδή υπάρχει είτε πλειοψηφία είτε συνασπισμό στο κοινοβούλιο. Α δούμε τι γίνεται στη Γερμανία, στην Ιταλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Πολωνία ή αλλού. Το κοινοβούλιο είναι υποχρεωμένο να στηρίξει την κυβέρνηση, επειδή ακριβώ υπάρχουν πλειοψηφικοί μηχανισμοί στην κοινοβουλευτική οργάνωση. Οπότε τις περισσότερες φορές η διάκριση των εξουσιών γίνεται σε όφελος της εκτελεστικής εξουσίας, γιατί πρόκειται για πλειοψηφία όπου είναι ο επικεφαλής ε, του πλειοψηφικού κόμματος, που είναι και ο επικεφαλής της κυβέρνησης στις περισσότερες περιπτώσεις. Πού είμαστε λοιπόν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάπου στη μέση. Στη μέση ενός προεδρικού συστήματος, στη μέση ενός κοινοβουλευτικού συστήματος, ε, και ακόμα και μέσα λίγο σε αυτή τη λογική της υπηρεσίας του οργανισμού. Πάντως, όπως συμβαίνει στο προεδρικό σύστημα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικρίνει τη δράση της Κομισιόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να την διαλύσει, προσπαθεί να έχει όσο και μεγαλύτερη επιρροή απέναντι στην Επιτροπή με διάφορους τρόπους, αυτό που κάνουμε και σήμερα εδώ. Ο έλεγχος του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή σημαίνει ότι η Επιτροπή ε, πρέπει πάντα να αποδεικνύει ότι κάνει σωστά αυτά που κάνει. Το Κοινοβούλιο βέβαια δεν μπορεί να προχωρήσει σε κυρώσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πολιτικού λόγου. Σήμερα όμω υπάρχουν και στοιχεία τα οποία μα πλησιάζουν στο κοινοβουλευτικό σύστημα. Για παράδειγμα, πώ αποφασίζεται η σύνθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά τι ευρωεκλογέ και ανάλογα με τα αποτελέσματα των εκλογών αυτών, αποφασίζεται η Επιτροπή και υπάρχει μια πλειοψηφία ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ενισχύει την αυτονομία της, κάτι το οποίο δεν είχαμε στο παρελθόν. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις εκλογές και μέχρι το Δεκέμβριο του 2016 υπήρχε ένας ισχυρός συνασπισμός στήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι ενισχύθηκε η Επιτροπή και ιδιαίτερα ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι ο μόνος σύμφωνα με τις συνθήκες που εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη συνέχεια αποφασίζει για τα μέλη του σώματος των Επιτρόπων, για τους Επιτρόπους. Η Επιτροπή δεν μπορεί να προχωρήσει σε διαδικασίες που επηρεάζουν τον κοινοβουλευτισμό πρέπει να συνοείται συνεχώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Γιούνκερ, για παράδειγμα, κέρδισε μέσω τη διαδικασία των Spitzenkandidaten νέα κοινοβουλευτική νομιμότητα που του προσέφερε αυτονομία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αν ήθελα να είμαι λίγο πιο προκλητικό, θα έλεγα ότι η υπόθεση Σαλμάγερ δεν θα είχε ε, συμβεί ποτέ αν δεν υπήρξε η διαδικασία των Spitzenkandidaten, γιατί δεν θα μπορούσε να έχει αντισταθεί στην πίεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Επιτροπή. Οπότε αυτή η λογική των Spitzenkandidaten επηρέασε και τη δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο στην Επιτροπή. Εγώ θα έλεγα ότι ενισχύονται με τον τρόπο αυτό και τα δύο όργανα. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται πιο σημαντικό παράγοντα στην πολιτική ζωή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εκλογέ έχουν περισσότερο νόημα για του πολίτε σήμερα, γιατί έχουν συγκεκριμένε συνέπειε. Η Επιτροπή από την άλλη μεριά διαθέτει περισσότερη δημοκρατική νομιμότητα και όχι μόνο μία νομιμότητα βάσει των συνθήκων. Δεύτερον, ενισχύεται η δυνατότητα κοινοβουλευτικού ελέγχου στην Επιτροπή. Εδώ τα πράγματα παίζονται. Επηρεάζει περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το πρόγραμμα τη Επιτροπή. Υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση με την Επιτροπή και το είπε και η κυρία Πρέσο ότι υπάρχει δυνατότητα steering, δηλαδή είναι ένα έλεγχος ο οποίο κατευθύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ τα που πρέπει να πάει. Από την άλλη, υπάρχει περισσότερη αυτονομία στην Επιτροπή, όπω είπαμε, και δυνατότητα κυρώσεων από το Κοινοβούλιο στην Επιτροπή χάνει κάπω τη δύναμή τη. Τέσσερα σημεία θα έπρεπε να προσέξουμε τώρα όταν προβληματιζόμαστε για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Πρέπει να δούμε και όλο το πλαίσιο. Πρώτο, ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που ελέγχει και ετοιμάζει του στόχου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Είναι δύσκολο έτσι να εισακουστεί περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει εδώ πέρα αυτό που λέμε με ένα σατρουά, δηλαδή τρεις βρίσκονται μέσα σε αυτή τη σχέση. Έπειτα υπάρχει το νομοθετικό έργο. Εδώ βρισκόμαστε σε κλασικό κοινοβουλευτικό σύστημα, όπου υπάρχει πραγματική συνεργασία και διαπραγματεύσεις μεταξύ των διάφορων εξουσιών. Αυτή η μέθοδος εργασίας οδηγεί σε περισσότερο έλεγχο, επηρεάζει περισσότερο το Κοινοβούλιο, αλλά με διακριτικό τρόπο. Και δύσκολα θα εξηγήσει στους εκλογείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα πού δραστηριοποιήθηκε στον έλεγχο αυτό, γιατί δεν είναι τόσο ορατό επικεντρώνεται στις νομοθετικές του δραστηριότητες και πιστεύω και ότι ο τριμερής διάλογος που ισχύει αποδυναμώνει το κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τρίτον, με ποιο τρόπο χρησιμοποιείται ο έλεγχος στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρησιμεύει για πολλά πράγματα φυσικά. Ε, συζητιέται η πολιτική της Επιτροπής, ε, την περιορίζει σε επιλογές της. Ναι, αλλά χρησιμεύει επίσης για κάποιους ευρωβουλευτές για να αντιτίθενται και να αντιπαρατίθενται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμεύει για κάποιου ευρωβουλευτέ επίση για να ακούγονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κυρίω αυτοί οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν εκθέσει και να προβληθούν μέσω αυτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολλέ φορέ αναγκάστηκε να περιορίσει τον έλεγχο γιατί η χρήση του ήταν καταχρηστική και δεν είχε τελικά και καμία σχέση με τον πραγματικό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και το τελευταίο που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μα αυτό τον προβληματισμό είναι η απομάκρυνση από την πολιτική. Εδώ πρέπει να επανέλθουμε στις αρχές του οικοδομήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αρχικός στόχος στη δεκαετία του 50 ήταν με τρόπο πλουραλιστικό και βάση πραγματογνωμοσύνης να αποφύγουμε την πολιτική στα πράγματα που δεν ήταν πολιτικά. Και ακριβώς και δημιουργήθηκε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτό το κεντρικό ρόλο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η απόσταση από την πολιτική είναι το μέσο για να λύσουμε τα προβλήματα. Όταν υπάρχει ένα σκάνδαλο, τι κάνουμε, μια υπηρεσία. Έχουμε τις τρελές αγελάδες, κάνουμε ε, μια υπηρεσία. Όταν είχαμε την κρίση της Ευρωζώνης, το διακανονίσαμε απομακρυνόμενοι από την πολιτική, δημιουργώντας τεχνικούς και τεχνοκρατικούς μηχανισμούς για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την υπόθεση. Το πρόβλημα είναι ότι όταν απομακρυνόμαστε από την πολιτική, απομακρυνόμαστε και από τον πολιτικό έλεγχο, γιατί η Ευρωπαϊκή θα πει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μα μη με επρίσετε, εγώ βάσει της πραγματογνωμοσύνης που διαθέτω παίρνω τις καλύτερες δυνατόν αποφάσεις. Και εδώ ο πρόεδρος Γιούνκερ δεν έχει σαφή τοποθέτηση. Και γι' αυτό πρέπει να ρωτηθούμε για αυτή τη διαδικασία το σπίτσε κατητάτεν. Είπε ο Γιούνκερ ότι ήθελε να είναι ένας πολιτικός πρόεδρος. Παρουσίασε ένα πολιτικό πρόγραμμα, μίλησε για την αρχή της πολιτικής ασυνέχειας και εδώ βασίστηκε στη γερμανική παράδοση που δεν υπήρχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε οι πρωτοβουλίε τη ε, Επιτροπή Μπαρόσο 2 δεν μα δεσμεύουν. Εμεί είμαστε πολιτική επιτροπή και θα τα κάνουμε αλλιώ. Συγχρόνω όμω όρισε το Φραν Τίμερμαν πρώτο αντιπρόεδρο, ο οποίο ασχολήθηκε με τη διαδικασία τη καλύτερη νομοθέτηση και ο ε, αντιπρόεδρο ε, Τίμερμαν είπε: Εμεί δεν κάνουμε πολιτική, κάνουμε επιστήμη. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να μπούμε στην ίδια λογική της πραγματογνωμοσύνης, στην οποία δεν μπαίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Πόψεβα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και ε, την κυρία Πρέσο και τον συγητή για την πρόσκληση. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα μιας μελέτης που έκανα για ένα βιβλίο, ε, το, του οποίου συντάκτης ήταν ο Λιβιέ Κώστα. Θα... Ήθελα λοιπόν ε, να σας παρουσιάσω το κεφάλαιο στο οποίο επικεντρώνομαι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Καταρχάς ε, λοιπόν θα πρέπει να καταλάβουμε την συνταγματική σημασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου και να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στον ε, έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας. Ε, ε, ο έλεγχος αυτός θεσπίζει την άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας για να έχουμε μια συνεχή αλυσίδα ευθύνης. Στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και ο καθηγητής Κώστα ήδη ανέφερε αυτές, αυτές ε, τις ε, αμφίσιμες έννοιες, διότι ποιος παίρνει τις αποφάσεις για να είναι δημοκρατικά νομιμοποιημένη η απόφαση. Χρειάζεται λοιπόν ε, να είναι θεμητές διαδικασίες. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στην ε, εκλογή του ε, κορυφαίου υποψηφίου, του Spitzenkandidat. Η νομιμοποίηση του αποτελέσματος γίνεται με βάση την ε, αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας για να διασφαλιστεί ένας ε, αντικειμενικός, μη πολιτικός έλεγχος της εφαρμογής. Αυτό λοιπόν αποτελεί σημαντική πρόκληση, το ότι έχουμε αυτή την αντίφαση όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ποιε είναι λοιπόν οι προκλήσει στον τομέα αυτών. Καταρχά, ποιο ελέγχεται. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε μια θεσμική ε, και όχι λειτουργική δηλαδή προσέγγιση ε, που έχουμε στα κράτη-μέλη. Ε, θα εξετάσω τα διάφορα μέσα του κλασικού ελέγχου Πάντω, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, ε, ο έλεγχο καλύπτει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι όμως μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εφαρμόζει και εκτελεί το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έχουμε λοιπόν ε, μία κάθετη δομή, έχουμε κατακαιρματισμό. Διότι και τα κράτη-μέλη ασκούν εκτελεστικές εξουσίες σε περιφερειακές αρχές και ιδιαίτερα στα ομοσπονδιακά κράτη-μέλη. Αυτό λοιπόν το πολυεπίπεδο σύστημα καθιστά δύσκολο τον αποτελεσματικό έλεγχο εάν εστιάζουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε οριζόντιο επίπεδο υπάρχουν διάφορες εκτελεστικές εξουσίες που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε κάποιες περιπτώσεις και στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή την είπα, εκπρόσωπο. και το Συμβούλιο ε, αλλά και οι Κομισιόν ε, μερικές φορές ασκούν εξουσίες που δεν τους έχουν δοθεί μέσω των συνθήκων. Δεν έχουμε μια έννοια εκτελεστική διαδικασία στις ε, συνθήκες, ούτε υπάρχει κατάλογος τομέων πολιτικής όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει αποκλειστική αρμοδιότητα. Πρόσφατα δε έχουμε και εκτελεστική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, για παράδειγμα, οικονομική διακυβέρνηση, ε, μέτρα κατά της οικονομικής κρίσης ε, κλπ. Αυτό είναι σημαντικό διότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή τα κράτη-μέλη διακυβερνητικά είπαν ότι εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι Ε, ο φορέας που ασκεί τέτοιες ε, εξουσίες οι οποίες ε, δεν απορρέουν από τη συνθήκη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να ελέγχεται από το Κοινοβούλιο. Πώς θα ασκείται λοιπόν αυτός ο δημοκρατικός έλεγχος για να είναι αποτελεσματικός. Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της δημοκρατίας, της συνένεσης Όλες οι αποφάσεις ε, θα πρέπει να γίνονται με βάση τη συνένεση. Πολλά παζάρια γίνονται, διαμεσολάβηση υπάρχει, ε, ε, συμβιβασμοί μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Είναι λοιπόν δύσκολο να εφαρμοστεί αυτή η ελεγκτική εξουσία του Κοινοβουλίου που ουσιαστικά διότι ουσιαστικά έχουμε εδώ πέρα δύο ανταγωνιστικά μεταξύ τους ε, θεσμικά όργανα, το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν ε, αποφάσεις λαμβάνονται σε πολύ πρώιμο στάδιο, όχι δηλαδή κατά την νομοθετική φάση, τότε είναι και πολύ δύσκολο για το Κοινοβούλιο να ελέγξει τις αποφάσεις αυτές εκ των υστέρων. Για να σας δείξω πώς αντικατοπτρίζονται οι προκλήσεις αυτές ε, στον σχεδιασμό των εργαλείων ελέγχου που έχουμε. Για παράδειγμα, ε, για παράδειγμα την πρόταση μορφή, ε, μπορεί, αυτό, μπορεί αυτή η πρόταση μομφής να έχει να κάνει με εκτελεστικές ε, δράσεις. Ε, εν τω μεταξύ, έχουμε πολύ ε, δραστικά μέτρα κυρώσεων, τα οποία όμως για να είναι αποτελεσματικά πρέπει να έχουν πολύ υψηλό κατόφλι. Μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ήταν πολύ πιο προσνής απέναντι σε ένα κοινοβούλιο που να έχει εκλεγεί μέσω αυτής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, θα ανταποκρινόταν πολύ περισσότερο απέναντι στα αιτήματα του Κοινοβουλίου. Επίσης, έχουμε την δυνατότητα ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ έχουμε και τις εθνικές αρχές, το οποίο είναι πολύ πιο ενδιαφέρον, διότι δεν καλύπτεται μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνεται υπόψη και το γεγονός ότι η εφαρμογή γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν έχει την δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, το Κοινοβούλιο μάλλον, να εξετάζει και τις εθνικές αρχές. Το πρόβλημα εδώ πέρα ε, είναι η συμμόρφωση με τα αιτήματα και τις συστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί ε, να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των σχετικών επιτροπών, όχι όμως τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη είναι μάλλον διστακτικά απέναντι σε τέτοια αιτήματα. Ε, έχουμε τον ε, κοινοβουλευτικό έλεγχο εκτελεστικών πράξεων. που ουσιαστικά θεσπίζουν δίκαιο. Και λέμε ότι εάν η εφαρμογή γίνεται από τις εθνικές ε, αρχές, ότι γενικά εφαρμόζεται από τις εθνικές αρχές, ποιος ελέγχει λοιπόν τις εκτελεστικές αυτές πράξεις. Ε, οι έρευνες δείχνουν ότι 50 με 60% όλων ε, των εκτελεστικών δράσεων σε Ευρωπαϊκή, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνονται με βάση εκτελεστικές πράξεις. Ποιο τα ελέγχει αυτά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να ελέγχουν μόνο ούλτραβύρες. Μπορούν δηλαδή μόνο να πούν ότι αυτή η εκτελεστική πράξη ε, ξεπερνά τις εξουσίες που δίδονται στην ε, βασική νομική πράξη, ενώ τα κράτη-μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τις εκτελεστικές πράξεις, ακολουθώντας τη λογική ότι αυτά είναι ουσιαστικά αρμόδια για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Και αυτό γίνεται μέσω της συμβουλευτικής διαδικασίας και της διαδικασίας ελέγχου, της νέας ε, διαδικασίας επιτροπολογίας δηλαδή. Εδώ όμως δεν έχουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο διότι στις επιτροπές αυτές ε, συμμετέχουν ε, αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων. Δεν υπάρχει εδώ λοιπόν κοινοβουλευτικός έλεγχος. Και όπως ανέφερα στο πλαίσιο του άρθρου 291 υπάρχει αυτή η εξουσία του Συμβουλίου να υιοθετεί εκτελεστικές πράξεις σε περιπτώσεις εφαρμοστικές πράξεις Ε, σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά πάλι ποιος ελέγχει το, ε, το Συμβούλιο στις περιπτώσεις αυτές. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Τα κράτη-μέλη λένε ότι τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να ελέγχουν τους εκπροσώπους τους σε αυτές τις επιτροπές. μπορούν να ελέγχουν ε, το πώς ε, διαμορφώνεται η πράξη αυτή, δεν μπορούν να ελέγξουν όμως το αποτέλεσμα. Ε, οι πανεπιστημιακοί λοιπόν αμφισβητούν όσον αφορά την δυνατότητα αυτή, την μη ύπαρξη μάλλον της δυνατότητας ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά έχουμε κάποια κλασικά μέσα για τον ε, τιμωρητικό εκ των υστέρων έλεγχο. Και εδώ πάλι το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι δεν έχουμε δυνατότητα στη συνθήκη για γραπτή ε, απάντηση ε, από το, από το Συμβούλιο. Αυτό επιτρέπεται μόνο στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ. Υπάρχει στον ε, κανονισμό η διαδικασία για τις ερωτήσεις, ε, δεν θεσπίζεται όμως στη συνθήκη. Ο πρόεδρος ε, Χέρμαν Φαν Ρόμποϊ, που ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου το 2010, δέχτηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις του Κοινοβουλίου για τις δικές του όμως πολιτικές δραστηριότητες, όχι για το Συμβούλιο. Αυτό που είναι ενδιαφέρον όσον αφορά τις γραπτές και προφορικές ερωτήσεις, και τον χρόνο ερωτήσεων είναι ότι είναι ad hoc. Δεν υπάρχει κατόφλι και ε, συνήθως χρησιμοποιούνται από μια κοινοβουλευτική μειοψηφία. Αν ε, λοιπόν ε, επιμείνουμε στις ε, πιο στενές πολιτικές σχέσεις ανάμεσα στο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τέτοια εργαλεία Τη μειοψηφίας θα λάβουν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Συνοψίζοντας, ε, ποια θα είναι οι λύσεις στα προβλήματα όσον αφορά τον έλεγχο. Όλες οι εκτελεστικές εξουσίες ε, θα πρέπει να ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υπάρχει δηλαδή ε, ένας ενιαίος εκτελεστικός φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σαφείς αρμοδιότητες εκτελεστικές. Έτσι, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος θα γίνει πολύ πιο αποτελεσματικός. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι θα χρειαστεί να αλλάξουμε ε, τον τρόπο λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πολύ συνένετικό. Αυτό ε, σχετίζεται και με τον κύκλο ε, την κατάρτιση των θεματολογίων κλπ. Ακόμα λοιπόν και αν όλες οι εκτελεστικές εξουσίες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρόλα αυτά θα είναι δύσκολο να ασκείται αποτελεσματικά ο έλεγχος. Δεν είναι κάτι νέο αυτό. Το Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια το κάνει αυτό, δηλαδή με τον ε, έλεγχο, τον εκ των προτέρων ε, έλεγχο προσπαθεί να αντισταθμίσει της ε, λήψης των κλασικών ε, μέσων που έχει στη διάθεσή του. Μαθαίνει δηλαδή από τις διαδικασίες και τις ενσωματώνει στις νέε προτάσεις. Και θα κλείσω εδώ με κάποια παραδείγματα σχετικά με τα εργαλεία αυτού του ε, κατευθυντικού ελέγχου, του εκ των προτέρων ελέγχου. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών προτεραιοτήτων, ουσιαστικά δηλαδή η κατάρτιση των θεματολογίων, κάτι που γίνεται με διάφορες διαδικασίες. Το Κοινοβούλιο το κάνει αυτό στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν, έχουμε την συζήτηση για την κατάσταση της Ένωσης και ε, μετά την ε, συμφωνία του 2016 για την καλύτερη νομοθεσία έχουμε και την ε, κοινή δήλωση σχετικά με τον διαθεσμικό προγραμματισμό. Αυτοί λοιπόν είναι τρόποι που βοηθούν το Κοινοβούλιο να συνδιαμορφώνει την ε, ημερήσια ε, διάταξη, τις προτεραιότητες ε, του θεματολογίου. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Κατόπιν έχουμε τις μελέτες αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Λιβιέ αναφέρθηκε στο πρόβλημα της διαμόρφωσης πολιτικής ε, με βάση ε, τεκμηριωμένα στοιχεία. Το πρόβλημα εδώ είναι φυσικά και ο Λιβιέ ε, το ανέφερε αυτό. Όποτε έχουμε μια τεχνική λύση που προβάλλεται ως η καλύτερη, πάντα συνεπάγεται μια πολιτική επιλογή. Και πολλές από τις μελέτες αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μπορεί να υπάρχουν διάφορε μελέτε αντικτύπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιλέγεται ε, μία η οποία μπορεί τεχνικά να είναι η καλύτερη, πολιτικά όμω να μην ενδείχνεται. Και γι' αυτό το Κοινοβούλιο άρχισε να εξετάζει τι μελέτε αντικτύπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δει αν οι λύσει που προτείνονται είναι πράγματι οι καλύτερε. Και έτσι να διατηρήσει την πολιτική επιλογή τελικά. Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνει αυτό και να μην ε, ε, βασιζόμαστε αποκλειστικά στον εκ έλεγχο. Επίσης, ε, εκθέσεις ε, εφαρμογής που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει ε, να δίνονται πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Αυτά λοιπόν είναι κλασικά εργαλεία ελέγχου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, το EPRS τώρα θα μιλήσει. Όσο πιο σύντομος ε, μπορείτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι συντομότατος. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την συγγήτρια της κυρίας Μπρεσό που ζήτησε από την Υπηρεσία Μελετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αναλάβουμε τη μελέτη και την ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που μας έδωσε κατά τη διάρκεια της έρευνας. Τα βασικά θέματα, μεθοδολογία και τα συμπεράσματα θέλω να αναφέρω. Παρουσιάζω μια μελέτη. Κοινοβουλευτικό έλεγχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφαρμογή των διατάξεων τη συνθήκη είναι ο τίτλο. Ο τίτλο ο ίδιο περιορίζει κατά κάποιο τρόπο την μελέτη. Επικεντρωθήκαμε μόνο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη μελέτη μα και των διατάξεων των συνθήκων. Η μελέτη ανετέθη τον Ιούλιο του 2018 και το όριο ετέθη από κάποιους περιορισμούς, τρεις στον αριθμό. Μεθοδολογικοί περιορισμοί καταρχάς. Εξετάζουμε συγκεκριμένες πράξεις, εφαρμογή της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν αυτού, πέρα από τις νομικές διατάξεις των συνθήκων, εξετάσαμε και άλλα έγγραφα νομικού χαρακτήρα, παρομφερή χαρακτήρα όπως των συνθήκων και συμπελήθησαν στην ανάλυση. Διοργανικές συμφωνίες, καλύτερη νομοθεσία για το 2016, η συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ένα άλλο έγγραφο, και διαδικαστικά στοιχεία εξετάσαμε, εσωτερικός κανονισμός του Ευρωκοινοβουλίου. Σε κάποια τμήματα της μελέτης μας εξετάζουμε και άλλα έγγραφα διοργανική συμφωνία για δημοσιονομική πειθαρχία, Φερρυπίν. Δεύτερος περιορισμός όσον αφορά την μελέτη. Αξιολογούμε μόνο τα όσα συνέβησαν με τέθεση ισχύ τη συνθήκη της Λισαβόνας. Από το Δεκέμβριο δηλαδή 2009 και πέρα. Εξ αυτού να μην θεωρηθεί το έγγραφο ότι είναι ιστορική μελέτη αλλά αξιολόγηση πραγματικών στοιχείων όσον αφορά την καθεστοιχεία τάξη τη σημερινή. Δίνουμε ποσοτικά στοιχεία και κάποια ποιοτικά, μάλλον ποιοτικά στοιχεία βασικά που στηρίζονται και από ποσοτικά. Σε κάποιες περιπτώσεις εξετάζουμε και ζητήματα που εντοπίστηκαν πριν το 2009. Στοιχεία που αναφέρονται για να δείξουμε ποια ήταν η πρώτερη πρακτική. Τρίτος μεθοδολογικός περιορισμός έχει σχέση με κάποιους τομείς. Εκεί που το Κοινοβούλιο έχει αρμοδιότητα ελέγχου. Επειδή είχαν περιορισμένο χρόνο για τη μελέτη, σε σύμφωνη γνώμη με, τον, με την εισηγήτρια, επικοινωθήκαμε βιδεκά των θεμάτων, εκλογικά θέματα, θέματα απόσυρση ψήφου εμπιστοσύνη, κυρώσει, απόσυρση ψήφου εμπιστοσύνη από επιτρόπου κλπ. Βασικέ πηγέ των στοιχείων. σε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες. Δημοσιεύματα στο σελίδα του Ευρωκοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και πιο σημαντική πηγή, οι πληροφορίες που λάβαμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ευρωκοινοβουλίου. Από όλε τι γενικέ διευθύνσει του Κοινοβουλίου συλλέξαν πληροφορίε. Presidency, IPOL, Φερρυπίν, Expo, και την νομική υπηρεσία. Και ευχαριστώ μάλιστα αυτές τις υπηρεσίες, τις γενικές διευθύνσεις που έδωσαν στοιχεία και που συνεργάστηκαν για τη μελέτη. Στα συμπεράσματα, αξιολογήσαμε την εφαρμογή των διατάξεων των συνθήκων εν συγκρίση με ευρύτερα κριτήρια. Πρώτο κριτήριο, ένταση των δράσεων του Κοινοβουλίου. Δεύτερον, συνέπειε, αντίκτυπο των δράσεων του Κοινοβουλίου, ένταση των δράσεων του Κοινοβουλίου, πόσο συχνά το Κοινοβούλιο χρησιμοποίησε τα προνόμια του όσον αφορά τον έλεγχο από το 2009 μέχρι το 2018. Πόσο συχνά δραστηριοποιήθηκε. Δεύτερον, αξιολόγηση αποτελεσμάτων. Ποια ήταν η αντίδραση Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τι ε, τις περιπτώσεις που άσκησε τα προνόμια του το Κοινοβούλιο είχαμε χαμηλή ένταση μέχρι υψηλή ένταση. Αυτή ήταν βαθμολόγηση. Χαμηλή ένταση δεν σημαίνει ότι ήταν επαρκή η δράση του Κοινοβουλίου. Έπρεπε να δούμε ότι κάποια προνόμια του Κοινοβουλίου είναι περιορισμένα χρονικά, όπω εκλογικά ζητήματα. Σε άλλα προνόμια του και δικαιώματά του, όπω οι νομοθετικέ διαδικασίε και η κατεξουσιοδότηση πράξη, σχετίζεται το όριο με την τεκμηριωμένη ε, γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Σε κάποιε περιπτώσει δεν κάναμε αξιολόγηση, δεν είχαμε αρκετέ πληροφορίε σε περιπτώσεις μικρών περιπτώσεων, μικρής ανάγκης παρέμβασης ή αν κάποιο προνόμιο δεν χρησιμοποιήθηκε για κάποια χρονική περίοδο όπως η ώρα των ερωτήσεων. Αντίθετα, η έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν κάποια όρια όσον αφορά τα αποτελέσματα ασκήσεως των προνομίων του Κοινοβουλίου έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάποιες τομείς. Και σε κάποιες περιπτώσεις που τίθενται όρια στα προνόμια από τις συνθήκες. Άρα δεν μπορεί να επηρεάσει πολύ τον αντίκτυπο το κοινοβούλιο. Δεν συμπεράναμε ότι οι δράσεις του κοινοβουλίου είναι χαμηλής έντασης, όμως σε κάποιες τομείς ίσως απαιτείται μεγαλύτερη προσοχή από το Ευρωκοινοβούλιο η πολιτική συζήτηση μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και άλλων θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Παράδειγμα, υιοθέτηση κανονισμού για το, για δικαίωμα του Κοινοβουλίου στην έρευνα. Κάποια συμπεράσματα, για να τονίσω κάποια πορίσματα. Αρκετά από τα προνόμια ελέγχου του Κοινοβουλίου είναι χρήσιμα σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είναι εκλογές που είναι χρονικά περιορισμένες ή ακροάσεις. Και αυτό επηρεάζει τα αποτελέσματα της ασκήσεως των δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου. Υπάρχει χρονικός περιορισμός αρκετά προνόμια ελέγχου που περιορίζονται χρονικά δεν χρησιμοποιήθηκαν εκτεταμένα ή καθόλου, όπως η δυνατότητα να ζητηθεί απόσυρση εμπιστοσύνης από κάποιον συγκεκριμένο επίτροπο. Ε, τρίτον, υπάρχει υψηλό όριο στο, στο, στην Ολομέλεια για τα προνόμια ελέγχου και αυτό εμποδίζει την άσκηση του ελέγχου. Όπως η πρόταση μομφής και μια επιτυχής άσκηση τέτοιου ελέγχου απαιτεί στενή συνεργασία όλων των πολιτικών ομάδων. Κλείνοντας, αναφέρω το τελευταίο σχόλιο ότι οι ειδικέ επιτροπές έρευνας και επιτροπές έρευνας δεν έχουν το δικαίωμα να καλέσουν μάρτυρες επίσημα ή να καλέσουν άτομα να υποβάλουν συγκεκριμένα έγγραφα. Και οπότε μειώνεται έτσι η πειθό, αν θέλετε, των ε, επιτροπών αυτών. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και όλους τους, ε, όλες οι υπηρεσίες που μας βοήθησαν και συνέβαλαν στην, με την υποβολή ε, πληροφοριών και μας βοήθησαν. Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις. Έχουμε ένα δεκάλεπτο για συζήτηση και να αφήσουμε και πέντε λεπτά για να απαντήσουν ε, οι συγκεκριμένοι. Ο Ραμόν Χαουρέγγι ήταν ο πρώτος. Μετά έχουμε τον Ρίτσαρντ, τον Έλμαρ και τον κύριο Βιασντόφσκι. Ο Ραμόν ήταν πρώτος. Θα συνοψίσετε, θέλετε να ξεκινήσετε εσεί, κυρία Μπεσό. Α, το τέλο καλύτερα. Ο Ραμόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ καταρχάς ε, του εμπειρογνώμονε και έχω δύο σχόλια όσον αφορά τις ελεκτικές εξουσίες του Κοινοβουλίου. Καταρχάς όσον αφορά τις επιτροπές ε, ε τις ερευνητικές. Εγώ πέντε χρόνια πέρασα ε, διαπραγματευόμενος με το Συμβούλιο και την, Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις εξουσίες που έχει μια Επιτροπή Έρευνας. Επιτροπή Ελέγχου. Παρά το άρθρο 227 των συνθήκων, παρά τα όσα επιτάσσει, που μπορεί να ασκήσει πειθαρχική εξουσία το Κοινοβούλιο, δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα κατάλληλο κοινοβουλευτικής δυνατότητας ελέγχου και τι εξουσίες έχουν οι ερευνητικέ επιτροπές. Και τελικά δεν δέχεται δεν δέχεται να, να ε, έχουν δυνατότητα επιτροπές, να έχουν το δικαίωμα να καλέσουν ε, μάρτυρες να ε, καταθέσουν. Δεν είναι ξεκάθαρες οι εξουσίες λοιπόν. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Διότι δεν εφαρμόζουμε πρακτικά τις συνθήκες που επιτρέπουν τη σύσταση και τη λειτουργία αυτών των επιτροπών των ερευνητικών. Είναι ένας μηχανισμός που είναι απαραίτητος για να γίνεται ο σωστός έλεγχος. Λοιπόν, καμιά φορά υπάρχουν λόγοι για να δημιουργηθεί μια ειδική ερευνητική επιτροπή, όπως στην περίπτωση των εγγράφων του Παναμά. Το πρόβλημα, τα σκάνδαλα του Λουξεμβούργου. η ασθένεια των τρελών αγελάδων. Όπου εκεί απαιτείται να έχει την εξουσία το Κοινοβούλιο, αλλά με τα σας λέω ότι ούτε το Συμβούλιο, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουν ε, να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πραγματικά αυτή τη δυνατότητα. Αναφέρομαι τώρα στις συνθήκες. Άρθρο 234. Το άρθρο 234 καλύπτει το δικαίωμα για πρόταση μομφής ε, κατά όλη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνολικά. Είναι μια ψήφο ε, μη εμπιστοσύνη, ούτω είπε. Το Συμβούλιο, αν παραστεί αναγκαίο, θα πρέπει να προτείνει τη σύσταση μιας νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Κοινοβούλιο. Δεν είναι η ίδια στάση όπως τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η έλλειψη όμως εφαρμογής του κανόνα για απόσυση ψήφου εμπιστοσύνης από συγκεκριμένο επίτροπο ε, εμποδίζει να ασκεί το δικαίωμά του για ψήφο μομφής, για πρόταση μομφής συλλογικά στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ τους τρεις εμπειρογνώμονες που πολύ σωστά μαζί παρουσίασαν τις διάφορες περίπλοκες πτυχές των διαφόρων στοιχείων και τι εξελίξει που είχαμε την πάρα του χρόνου. Η κατάσταση και το σύστημα δεν είναι στατικό. Είχαμε συνεχή εξέλιξη και έτσι θα συνεχιστεί. Ίσως με αυξανόμενους ρυθμούς και με κάποια μπλοκαρίσματα, όπως μας είπε και ο Ραμόν. Νομίζω με την πάροδο του χρόνου όμως θα ε, συνεχιστεί αυτή η εξέλιξη και οι αλλαγές. Κάποιες ανησυχίες εξεφράστησαν, εγώ δεν ανησυχώ τόσο. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι ένα τμήμα του εκτελεστικού κλάδου. Τι γίνεται με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή της ΥΠΑ εκπροσώπου ή άλλων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εντοπίζει στο, στατηγικές προτεραιότητες και θέτει επιτάπητος θέματα και καμιά φορά ανεβάζει θέματα από εθνικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά δεν είναι ο καθημερινός εκτελεστικός φορέας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το ευρωπαικο συμβουλιο εντοπιζει στο προτεραιοτητε προτεραιοτητες και θετει επιταπητος θεματα και καμια φορα ανεβαζει θεματα απο εθνικο σε ευρωπαικο επιπεδο αλλα δεν ειναι ο καθημερινος εκτελεστικος φορεας η ευρωπαικη επιτροπη εχει το προσωπικο που εφαρμόζει διάφορα μέτρα, έχει τον προπολογισμό και έχει να αντιμετωπίσει τι καθημερινέ εκτελεστικέ λειτουργίε. Και είπα ότι εκπρόσωπο στο κάτω-κάτω είναι αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίτροπο. Ο Χέρμαν Βαν Ρόμποϊ, πρώην πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είπε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι κινητήρια δύναμη, αλλά δεν είναι συνδεδεμένη, είναι μονάδα παραγωγή ενέργεια, δεν συνδέεται με το δίκτυο. Όταν είναι να εφαρμοστούν διάφορα πράγματα, άλλοι θεσμικοί φορεί να το κάνουν, άλλα θεσμικά όργανα. Αυτό δεν με προβληματίζει τόσο. Επίσης, δεν ανησυχώ για διάφορες λεπτομέρειες που αφορούν τις ελεγκτικές μας δυνατότητες. Έχουμε ένα φάσμα αυτών που έχουν αυξηθεί. Δεν ανησυχώ τόσο πολύ ότι χρησιμοποίησαμε μόνο την ψήφο μορφή μία φορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τεχνικός πώς δεν το κάναμε καν αυτό, παρετήθηκε πριν ψηφίσουμε. Το γεγονό ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε κοινοβούλιο καθιστά σαφέ ότι ο εκτελεστικό κλάδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προσέξει το κοινοβούλιο, όπω και τα εθνικά κοινοβούλια. Είναι ασυνήθιστο να υιοθετήσουν ψήφο μία απόσταση εμπιστοσύνη από την κυβέρνηση. Μία φορά συνέβη στη χώρα μου, μόνο μία φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γεγονό ότι μπορεί αυτό να συμβεί δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα λογοδοσία και αν τα όρια. Υπάρχει δημοκρατία, δύνασε να το πράξεις και η κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί με κάποια προσοχή. Είναι η αρχή ε, της κρυφής δύναμης, των κρυφών ε, ε, εξουσιών, των κεκαλυμμένων. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τις χρησιμοποιήσεις πάντα, αλλά το ότι μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις είναι σημαντικό. Ούτε με προβληματίζει ότι μια ψήφος μομφής, μια πρόταση μομφής δεν δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να διαλύσει ε, κοινοβούλιο, το κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόορες εκλογές. Στη Νορβηγία δεν μπορούν να προκηρυχθούν πρόορες εκλογές, ούτε στην Ελβετία και στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει πολύ πιο δύσκολο αυτό. Με ένα νόμο για σταθερή θητή του Κοινοβουλίου και στη Γερμανία πολύ δύσκολο μια φορά να συνέβη στην ιστορία. Αλλάζει την κυβέρνηση με άλλο τρόπο δεν χρειάζεται να προκηρυχθούν πρόορες εκλογές και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο νομίζω πιθανότατα ότι αυτό είναι και σοφό έτσι που στην κατάσταση που βρίσκεται η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αληθεύει, δεν έχουμε ειδικέ εξουσίες όσον αφορά τις εφαρμοστικές ε, ε, πράξεις. Δεν έχουμε συγκεκριμένες εξουσίες ελέγχου, αλλά εμπίπτουν στα πλαίσια των, γενικών μας δικαιωμάτων ελέγχου. Να υποβάλουμε ερωτήσεις, να καλέσουμε αξιωματούχου ε, των επιτρόπων να εξηγήσουν σε κοινοβουλευτικέ επιτροπές, να δικαιολογήσουν κάποιες πράξεις. Έχουμε το δικαίωμα να μπλοκάρουμε πληρωμέ για οποιαδήποτε εφαρμοστική ε, απόφαση που έχει επιπτώσει για τον προπολογισμό. Έχουμε διάφορους τρόπους, όχι αν συγκεκριμένο, σε εθνικές περιπτώσεις όπως στη Γαλλική. Έχει σημαντικό περιθώριο κυβέρνηση για να εφαρμόσει ρυθμιστικές εξουσίες που αποκαλούνται στη Γαλλία χωρίς κάποιο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εμείς έχουμε περισσότερες δυνατότητες από ότι κάποια εθνικά συστήματα μπορεί να βελτιωθεί. Αυτό θα βελτιωθεί σταδιακά, αλλά δεν νομίζω ότι είναι θεμελιώδες πρόβλημα ή αδυναμία. Τώρα για φιλοσοφικά ζητήματα. Αυτό που έθεσε ο κύριος Κώστα, η, τάση που, η ένταση που υπάρχει μεταξύ του ρόλου ενός τεχνικού φορέα και του, ενός πολιτικού φορέα την ίδια ένταση αυτή, την ίδια ένταση μπορείς να την δεις διαφορετικά. Την ένταση μεταξύ συνενετικής πολιτικής και πολιτικής που ασκείται μέσω της πλειοψηφίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υβριδικής μορφής, διότι η Ένωση 28 διαφορετικών χωρών, μέρη για αυτό το λόγο. Αλλά έχουμε αποφάσεις που λαμβάνονται συνενετικά στο Συμβούλιο, όπου χρειάζεται ειδική πλειοψηφία και είναι υψηλό όριο, δεν είναι απλή πλειοψηφία. Και σε κάποια πράγματα χρειάζεσαι και ομοφωνία. Στο κοινοβούλιο όμω έχουμε πλειοψηφίε. Απλή πλειοψηφία. Συνήθω. Συνήθω, όχι πάντα. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα κολέγιο, ένα φορέα που πολιτικό πώ είναι μια μόνιμη συμμαχία. Πάντα υπάρχουν σοσιαλιστέ, ΕΛΚ, φιλελεύθεροι και καμιά φορά και άλλοι που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν διαμορφώνεται κάποια πλειοψηφία. Είναι κάτι σαν την ελβετική κυβέρνηση που αποτελείται από μόνιμη συμμαχία των ίδιων τεσσάρων κομμάτων, από ό,τι θυμάται κάποιο. Ό,τι και να γίνεται σε εκλογέ. Πάντα τα ίδια κόμματα. Είναι συνενετική η προσέγγιση. Αλλά με το σύστημα candidaten πήγαμε σε μια επιλογή ε, επιβολής πλειοψηφία. σε σημαντικό βαθμό. Όσον αφορά τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε υβριδικό σύστημα. Έχουμε το ελβετικό συνενετικό σύστημα και το σύστημα το πλειοψηφικό ή τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως και το σύστημα γενικά έχουμε συνενετική πολιτική στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο σε, μεγάλο βαθμό και το σύστημα της πλειοψηφίας στο Ευρωκοινοβούλιο και προσπαθούμε να βρούμε ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών συστημάτων δοθήσεις καταστάσεως της παρούσης της Ευρωπαϊκής Ολοκληρώσεως Έχουμε ισχυρά κράτη με χαρακτήρα, εξουσίες και ιστορία και πολιτικά συστήματα, ίσως αυτή είναι σοφή ισορροπία. Μεταλλάσσεται, εξελίσσεται, κινούμεθα προς ένα σύστημα που χρησιμοποιεί όλο και πιο συχνά την πλειοψηφία, περισσότερες φορές χρησιμοποιεί η πλειοψηφία το Συμβούλιο, σπίτσαν κατηντάτεν, ισχυρότερε εξουσίες στο Κοινοβούλιο, αλλά ε, είναι υβριδικό το σύστημα ακόμα και θα εξακολουθεί να αλλάζει και να εξελίσσεται. Εγώ δεν θέλω να δραματοποιώ το γεγονός ότι είναι ε, υβριδικό το σύστημα. Ευχαριστώ, Ρίτσορτ. Έλμαρ Μπρόκ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ε, γνωρίζω κανένα δημοκρατικό σύστημα που να μην έχει τις ιδιαιτερότητες του. Νομίζω ότι ο καλύτερος έλεγχος ε, πραγματοποιείται όταν ε, η εκτελεστική εξουσία φοβάται. Πώς μπορεί όμως να οργανώσει κανείς το φόβο. Θα πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες ώστε να μπορεί κανείς ε, να το ελέγξει αυτό. Ε, είχαμε μία περίπτωση όπου η Κομισιόν ε, δεν μπόρεσε να τη γλιτώσει, αλλά πλειοψηφία των δύο τρίτων ε, δεν είναι αμεληταία. Δεύτερο σημαντικό θέμα είναι η διαδικασία του κορυφαίου υποψηφίου, του Spitzenkandidat, ε, να γίνεται από το Κοινοβούλιο. Έτσι θα έχουμε περισσότερη επιρροή από ότι πολλά εθνικά κοινοβούλια. Επειδή όμως ε, το Κοινοβούλιο δεν έχει μία μόνιμη κυβερνητική πλειοψηφία, ε, οι επίτροποι ε, πάντα προέρχονται από την μειοψηφία και αυτό λοιπόν είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι ένας ε, που εκλέγεται πρόεδρος της Επιτροπής ε, έχει ήδη προειδοποιηθεί επαρκώς. Πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε το θέμα της εφαρμογής της νομοθεσίας. Πάντα αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. αλλά δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά όσον αφορά την εφαρμογή. Ε, και στον τομέα αυτό έχει αποτύχει η συνθήκη της Λισαβόνας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα για να απαιτήσουμε ε, δικαιώματα ελέγχου που αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Εξετάζουμε δηλαδή αν έχουν δαπανηθεί σωστά οι πόροι. Αλλά δεν θα ήταν λογικό ένας εισηγητής και μετά την ε, έγκριση της έκθεσης να παραμείνει στο θέμα και μετά τρία-τέσσερα χρόνια να εξετάσει τι απέγινε η νομοθεσία αυτή. Δεν έχουμε καμία τέτοια εξουσία στο Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε εγκρίνει μια έκθεση, την ξεχνάμε. Δεν ε, έχει έλεγχο της εφαρμογής το Κοινοβούλιο. Εάν το είχαμε αυτό και είχαμε ε, τα δεδομένα μπροστά μας, θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε με πολύ περισσότερη ισχύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα λοιπόν του ελέγχου είναι θέμα κλειδί. Σε ένα ομοσπονδιακό σύστημα που η εφαρμογή βρίσκεται στα χέρια των κρατών μελών ή των περιφερειών. Κάτι που άλλο σωστό είναι σε ένα ομοσπονδιακό σύστημα. Αλλά εάν δεν υπάρχει έλεγχος, αυτό είναι πρόβλημα. Όσον αφορά ε, τους οικονομικούς πόρους, ε, γίνεται ο έλεγχος. Πρέπει λοιπόν να έχουμε και αυτό το δικαίωμα του ελέγχου και αυτό μπορούμε μόνο να το πετύχουμε εάν μπορούμε να έχουμε μάρτυρες ε, και να μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις μετά, να υποβάλλονται τα σχετικά έγγραφα και να υφίστανται οι ένοχοι όλες τις επιπτώσεις. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ βασικό πρόβλημα. Έτσι θα είχαμε μια σωστή ευκαιρία να πετύχουμε κάτι. Αλλά έχουμε αποτύχει μέχρι στιγμή στο θέμα αυτό και είναι κεντρικό όσον αφορά τις εξουσίες. Η εξουσία ελέγχου λοιπόν θα πρέπει να ενισχυθεί πολύ σε σχέση με το τι ήταν τα τελευταία 50 χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Κύριε Σουζαντόφσκι. Ευχαριστώ πολύ τους εμπειρογνώμονες για τις παρουσιάσεις τους. Έχω κάποιες ερωτήσεις στον καθηγητή Κώστα. Για τις άλλες, τις λοιπές πτυχές σχέση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής, εσείς αναφερθήκατε στην πτυχή έλεγχος. Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω την επιρροή κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πρόγραμμα της πολιτικής δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις νομοθετικές της προτάσεις. Πώς επηρεάζονται όλα αυτά. Υπάρχει ο έλεγχος, αλλά υπάρχει και η επιρροή της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στο πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μερσέντες τώρα Θέλετε το λόγο ή μετά τους εμπειρογνώμονες. Όπως θέλετε. Τώρα. Ωραία. Καλώς. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Θα περιοριστώ σε δύο λόγια μετά από αυτά που ακούσαμε και θα σας μεταφέρω και κάποιο προβληματισμό μου μετά από αυτά που είπε ο κύριος Κόρμπετ. Είναι αλήθεια ότι το σύστημα αυτό του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έλεγχο στην Επιτροπή και γενικότερα των πράξών της, εγγράφεται μεταξύ δύο πόλων του συνταγματικού ελβετικού ας πούμε. Η Ελβετία συνεχίζει με αυτό το σύστημα μη πλειοψηφικό στο μοσποδιακό σκέλος. Διότι σε μια τέτοια περίπλοκη περίπτωση όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση το να κρατήσουμε και αυτή την πτυχή που είναι πιο τεχνικός και πιο συνεντικός ίσως ε, να είναι κάτι πιο σημαντικό για τον έλεγχο όμως υπάρχει και άλλο στοιχείο που απορρέει από την πολιτική ιστορία των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών που στρεφόμαστε προς ένα έλεγχο πιο πολιτικής φύσης ε, την, υποστηρική, ε, την υποστήριξη στην πολιτική για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλη αυτή η διαδικασία του speech and candidate προς εκεί κινείται. Και οι δύο τρόποι του ελέγχου πιστεύω ότι είναι σημαντικοί, πρέπει να διατηρηθούν διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, ένα υβρι, είναι υβριδικής μορφής. Ίσως μια προσεχής αλλαγή των συνθηκών μπορεί να το λάβει καλύτερη υπόψη. Είναι δύο μοντέλα κάπως διαφορετικά που λίγο πολύ πρέπει να διαλέξουμε. Αν θα διαλέξουμε το σύστημα περισσότερο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως είναι προεδρικό το σύστημα, όπως είπε ο καθηγητής Κώστα, ή ένα μοντέλο πιο πολύ συμμετοχικό, όπου ο ρόλος των πλειοψηφιών και των μειοψηφιών είναι πιο ασθενής ή σχεδόν δεν υπάρχει. Εγώ θα έδινα όμως και σημασία στη δουλειά που θα κάνουμε, στον προβληματισμό που θα κάνουμε όσον αφορά το θέμα του κάθε του ελέγχου, που θεωρώ ότι είναι άλλο σημαντικό ε, στοιχείο σε ένα σύστημα ιονή ομοσπονδιακό, κάτι το οποίο δεν είμαστε ακόμα ομοσπονδιακό. Οι σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια, περιφερειακά κοινοβούλια, με το Ευρωκοινοβούλιο κάτι που χρειάζεται για να είναι αποτελεσματικότερος έλεγχος όσον αφορά το σύνολο των πράξεων που υθετούμε για να είμαστε πιο σίγουροι ότι στο τέλος τα αποτελέσματα υπάρχουν. Και αυτό πιστεύω ότι είναι προς συμφέρον και δικό μας και των Εθνικών και Περιφερειακών Κοινοβουλίων. Και τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τις εκκλήσεις που ακούστηκαν από τον καθηγητή Κώστα. Το να μεταφέρουμε, ε, να, να πάρουμε εξουσίες από τις διάφορες υπηρεσίες ή, ή μάλλον να στρεφόμεθα προς τεχνικούς φορείς είναι κάτι που δυσκολεύει τους ελέγχους. Και νομικά περιπλέκεται η κατάσταση διαφορετικό έλεγχο ενό τεχνικού φορέα από ότι ο έλεγχο επί ενό πολιτικού φορέα. Αλλά αναθέτουμε τελικά εξουσία στον τεχνικό φορέα πολιτική φύσεω. Και έτσι μπερδεύονται τα πράγματα και γίνονται πιο ανάμεικτα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε μόνο στα πλαίσια τη εκθέσεω. Πιθανότατα θα πρέπει αυτό είναι ένα αρμοδιότητα ε, που θα αναλάβει η επόμενη θητεία. Είναι πάρα πολύ περίπλοκο και όμως είναι θεμελιώδου σημασία να γίνει ένας προβληματισμός βλέποντας τον απίστευτο αριθμό μέσων υπηρεσιών που έχουμε αυτού του τύπου και που δημιουργήσαμε και που δημιουργούμε. Α, ευχαριστώ. Και να δώσουμε το λόγο στους εμπειρογνώμονές μας πάνω απ' όλα δεν έχετε όσο χρόνο θα θέλατε να έχετε, αυτό το ξέρετε, έτσι. Παρακαλώ, κύριε Κώστα. Ναι, θα είμαι σύντομος. Όσον αφορά τον έλεγχο, ο έλεγχος ε, βάζει προβλήματα στο Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα χρόνου για τους εκλεγμένους, αρμοδιότητας όταν είναι πολυτεχνικά τα θέματα, αλλά και διάθεση, γιατί κανένας ευρωβουλευτή δεν θέλει να κάθεται και να ξεφυλίζει την επιτροπολογία. Ε, ξέρει ότι κινδυνεύει να θαυτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάτω από τόνους χαρτιού. Το ίδιο ισχύει και στα εθνικά κοινοβούλια για την επικουρικότητα. Ελάχιστοι ευρωβουλευτέ έχουν την όρεξη να ασχοληθούν με αυτό ή ξέρουν. Οπότε είναι ζήτημα οργάνωσης επίσης. Εξού και τελικά πηγαίνει σε διοικητικές υπηρεσίες η αρμοδιότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου και το κοινοβούλιο απλώς εποπτεύει και συγκεντρώνει τα δεδομένα. Για την ερώτηση του Ευρωβουλευτή όσον αφορά την επιρροή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εγώ πιστεύω ότι ήταν αξιοσημείωτη στην αρχή της θητείας όταν έγιναν οι διαπραγματεύσεις με τον Κλοντ Γιούνκερ όσον αφορά το πρόγραμμα της θητείας και υπήρξε συμφωνία μεταξύ των σοσιαλιστών, των φιλελεύθερων και του ΕΛΚ για το Ταμείο Γιούγκερ. Εδώ η συνάδελφος έχει περισσότερα στοιχεία και πιο ουσιώδη, αλλά είναι ακριβώς η αδυναμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μπορέσει να εισακουστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο πρόεδρος ε, Ταγιάννη πήγε στο Κολέγιο της Ευρώπης στην αρχή της ακαδημαϊκής ε, χρονιάς και μίλησε για το δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα. Πολύ σύντομα να απαντήσω και εγώ στον κύριο Κόρμπετ πρώτα απ' όλα. Συμφωνώ μαζί σας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όντως ε, αναλαμβάνει αυτό πολλές από τις στρατηγικές αποφάσεις. Αυτό που θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι πώς αυτή η συνεχής προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ζητήσει από την Επιτροπή να βάλει πράγματα στην ημερήσια διάταξη μερικές φορές κρατάει μήνες η διαδικασία, πάρα πολύ χρόνο. Εκεί ίσως θα έπρεπε να υπάρξει περισσότερη ισορροπία μεταξύ των εξουσιών. Έπειτα για τον κάθετο έλεγχο, στον οποίο αναφέρθηκε η κυρία Μπρέσο. Συμφωνώ. Ακριβώς αυτή είναι η πτυχή που λείπει στο σύστημα του εκτελεστικού φεντεραλισμού. Μιλάμε πολύ για την αιρεσιμότητα στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, κονδυλίων δηλαδή που εκταμιεύονται ανάλογα με τις επιδόσεις. Σίγουρα υπάρχουν αδυναμίες στην ε, αποτελεσματικότητα της δίκησης. Και εγώ θα ήθελα πολύ σύντομα, επιτρέψτε μου, να αντιδράσω σε αυτά που ακούσαμε. Πρώτον, κάτι που είπε ο κύριος Μπροκ για το φόβο. Στην μελέτη μου, πολλές φορές αναφέρομαι, αν όχι στο φόβο, αν μη τι άλλο, στην απειλή του κοινοβουλευτικού ελέγχου και στα προνόμια που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα να πω και κάτι για τους πίτσεν τους επικρατέστερους υποψηφίους η διαδικασία αυτή χρησιμοποιήθηκε μία μόνο φορά. Τώρα θα είναι η δεύτερη. Και ήδη πριν από μερικές εβδομάδες ο πρόεδρος Τάσκ είπε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Συνεπώς, ναι, εδώ θα πρέπει να υπάρχει κάποια πολιτική συνεργασία, πολιτικές συζητήσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για διάφορα πράγματα, ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην τελικά απορρίπτει όλους τους υποψήφιους μέχρι να προταθεί αυτός που θα είναι ο Σπίτσε Κατιντάτ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Παρέβασε εκτός μικροφώνου της κυρίας Μπρέσο. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων αυτών και θα έλεγα και για να γραφτεί στα πρακτικά όταν έρθει το νέο κοινοβούλιο, στη νέα θητεία δηλαδή των συναδέρφων, να ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο όμως τελικά, που δεν υπογραμμίστηκε αρκετά, είναι το Συμβούλιο πώς συμμετέχει στον ετήσιο προγραμματισμό και ο έλεγχος ε, του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή, πώς επηρεάζεται από το χρονοδιάγραμμα. Όλα αυτά είναι προκλήσεις για μας. Ήταν μια πολύ καλή ακρόαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπορούσατε εσείς οι δύο ό,τι οι διαφάνειες ή ό,τι έχετε να μας τα δώσετε, να τα βάλουμε κι εμείς ε, στην ιστοσελίδα μας. Θα ήταν πολύ χρήσιμο και για τους συναδέρφους που δεν ήταν εδώ. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν και τους δυο σας και τον εκπρόσωπο του PRS. Και έτσι κλείνω το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη και περνάμε στην έκθεση Λαμασούρ. Εδώ πέρα πρόκειται για την εφαρμογή των διατάξεων των συνθήκων σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία. Έχουμε και εδώ δύο πυρογνώμονες. Ο πρώτος είναι ο Δόκτωρ Wolfgang Wessels από το Κέντρο Σπουδών για την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση από το Πανεπιστήμιο της Κολονίας και έχουμε και τον Κάρστεν Γκέραρτς από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Διπλωματικών Σπουδών, Κολέγιο της Ευρώπης. Θα κάνουμε μια εισαγωγή, κύριε Λαμασούρη, μετά να περάσουμε σε εμπειρογνώμονε. Παρακαλώ. Αλλά ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους δύο καθηγητές που έχουμε μαζί μας και τους ευχαριστώ και για το έγγραφο το οποίο μας έδωσαν και που θα σχολιάσουν βέβαια τώρα. Εγώ απλώς υπενθυμίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την επιθυμία να εκπονήσει μία έκθεση για την ενισχυμένη διαδικασία και την εφαρμογή της για να δούμε κατά πόσο από τις εμπειρίες που έχουμε συλλέξει μέχρι τώρα από βέβαια κάπου έξι περίπου ενισχυμένες διαδικασίες. Να δούμε λοιπόν κατά πόσο αυτή η διαδικασία μπορεί να χρησιμεύσει και σε άλλους τομείς ευρωπαϊκής πολιτικής επιμερισμένης αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών μελών για τις οποίες διαπιστώνουμε ότι κάποιες χώρες θέλουν να προχωρήσουν πιο γρήγορα προς κοινέ αποφάσεις, ενώ κάποιες άλλες δεν θέλουν να συμμετέχουν ακόμα. Αν αποδειχτεί αυτό, θα δούμε. Μήπως μπορούμε να έχουμε έτσι μια πιο καταστατική ενισχυμένη συνεργασία και να δούμε τι μπορεί να λυθεί με την ενισχυμένη συνεργασία. Οι συνθήκες, βλέπετε, δεν είναι αρκετά συγκεκριμένες για το πώς λειτουργεί. Ε, μιλάει για την προϋπόθεση βάσει της οποίας μπορούν να υπάρξουν τέτοιες ενισχυμένες συνεργασίες λέει σε ποια θέματα θα μπορούσε να υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία. Λέει τι πρέπει να γίνει με τις χώρες που δεν συμμετέχουν σε αυτήν, αλλά όσον αφορά τη λειτουργία της, με ποιο τρόπο λαμβάνονται οι αποφάσεις, ποια είναι η διοικητική οργάνωση, Ποιο είναι ο κοινοβουλευτικό έλεγχος, ο οικονομικός, η χρηματοδότηση κλπ. Η συνθήκη δεν λέει τίποτα. Γι' αυτό και θελήσαμε για να ετοιμάσουμε την έκθεση αυτή να ε, συμβουλευτούμε και να μάθουμε πρώτα απ' όλα τι συμβαίνει αλλού, στα ομοσπονδιακά δηλαδή συστήματα, όπου υπάρχουν διαδικασίες που επιτρέπουν στο εσωτερικό του ομοσπονδιακού συστήματος να υπάρχει συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επιπέδων, ακόμα και αν δεν συμμετέχουν όλα τα ομοσπονδιακά μέρη. Και από την άλλη θελήσαμε να έχουμε πραγματογνωμοσύνη, και αντικειμενική τοποθέτηση και αξιολόγηση όσον αφορά τις περιπτώσεις όπου μέχρι τώρα χρησιμοποιήθηκε αυτή η ενισχυμένη συνεργασία. Εξού και οργανώσαμε την ακρόαση για να ακούσουμε εκπροσώπους από τα διάφορα θεσμικά όργανα. Και σήμερα η ακρόασή μας προβλέπει την παρέμβαση ακαδημαϊκών που θα μας βοηθήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, αλλά. Ο καθηγητής Βέσελ πρώτα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές. Θα ήθελα ε, την εισαγωγή μου να την κάνω με τον τρόπο που ε, την κάνουμε πάντα στα πανεπιστήμια. Ερευνητές είμαστε, δεν έχουμε τις τελικές απαντήσεις, ε, πόσο μάλλον στη συγκεκριμένη περίπτωση. Νομίζω πολλοί από εμά εδώ έχουμε πολύχρονη πείρα με αυτά που μόλις ε, ανέφερες. Έχουμε ένα θεματολόγιο, θέλουμε να προχωρήσουμε με το θεματολόγιο αυτό και Ε, αναζητούν ε, πολλές χώρες ε, λοιπόν την επίλυση προβλημάτων με τις λεγόμενες υποομάδες. Δεν ξέρω αν θυμάστε την έκθεση Τίνερμανς για όσους έχουν μελετήσει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα θυμούνται ότι πρόκειται για ενδιαφέρουσα έκθεση για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητος όπου προέκυψαν ακριβώς τα προβλήματα αυτά, το δίλημα. Κάποιες χώρες να προχωρήσουν εντός ενός πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, χωρίς να είναι όλοι έτοιμοι ή διατεθειμένοι να ε, συμμετάσχουν σε αυτό το πλαίσιο ε, παράγοντας ταυτόχρονα δίκαιο το οποίο να μην αποτελεί μέρος του κοινοτικού κεκτημένου. Έχουμε λοιπόν από τη μία αυτούς που είναι υπέρ αυτών των υποομάδων και έχουμε και αυτούς που είναι υπέρ της ε, κοινοτικής ορθοδοξίας, ε, να το πούμε έτσι, και δεν τον εννοώ αρνητικά τον όρο αυτόν. Η πρόεδρος ε, και ο εισηγητής μας ζήτησαν να βρούμε ένα πρότυπο πλαίσιο. Αυτό νομίζω αναφέρατε. Θα θέλαμε να δούμε να βρούμε κανόνες και διαδικασίες που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους και γενικά και να μην χρειάζεται να τους εφεύρουμε κάθε φορά. Βλέπουμε εκτός του κοινοτικού πλαισίου ότι πολλοί επανεφεύρουν τον τροχό συνεχώς και νομίζω ότι το πιο χτυπητό παράδειγμα γι' αυτό είναι το Δημοσιονομικό Σύμφωνο που είναι ένας πολύ καλός τρόπος να είναι κανείς ευέλικτο, αλλά δεν ε, ανήκει στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωση. Τα ευρωπαϊκά όργανα, λοιπόν, με επικεφαλή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ελέγχονται από το δικαστήριο ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά ε, τα θεσμικά όργανα μπορεί να αποτελούν περιορισμό σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να δημιουργούν επιπλέον μπλοκάρισμα για κάποιες χώρες. Μία λοιπόν ε, ε, σύντομη επισκόπηση από μένα, μία σύντομη εισαγωγή για αυτά που θα σας πει ο συνάδελφος Κάρστεν. με τη συνθήκη του Άμστερνταμ είχαμε την ενισχυμένη συνεργασία, αλλά χρειάστηκε να οριμάσει επί πολύ καιρό μετά την ε, υιοθέτηση της συνθήκης της Λισαβόνας. Είχαμε πια χρήση της ενισχυμένης συνεργασίας. Ελάχιστες περιπτώσεις, ο Κάρστεν θα σας αναφέρει ποιες ήταν αυτές. Ενώ στο διάστημα αυτό βλέπουμε ταυτόχρονα ότι χρησιμοποιήθηκε η ευελιξία με διάφορους τρόπους ε, η αντιμετώπιση της ε, οικονομικής κρίσης ε, έγινε εκτός πλαισίου της συνθήκης και υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Είναι όμως πολύ σημαντικό. Επίσης υπάρχει πολύ χαμηλή ορατότητα της ενισχυμένης συνεργασίας και πολύ πιο επίκαιρο αυτή τη στιγμή είναι η ΠΕΣΚΟ, η μόνιμη συνεργασία και οι σχετικές διαδικασίες. Θα δούμε λοιπόν τι ε, συμπεράσματα μπορούμε να εξάγουμε από τη χρήση της μόνιμης διαθρωμένης συνεργασίας. Και ε, δύο ε, πτυχές θα σας παρουσιάσουμε τώρα, αφενός τον νομικό κόσμο και κατόπιν τον πραγματικό κόσμο. Α, δεν ολοκληρώσατε, λέει η πρόεδρος. ναι, παρακαλώ, συνεχίστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, πράγματι, έχουμε χωρίσει σε δύο τμήματα την ανάλυση μας. Έχουμε ε, τα νομικά λόγια, τον πραγματικό κόσμο και χρήσιμο είναι να αναφέρουμε ότι την μελέτη μας συμπληρώνει η εις μελέτη του EPRS σχετικά με, φορείς, με δομές διακυβέρνησης και τρόπους χρηματοδότησης. Στο... Καταρχάς λοιπόν επικεντρωνόμαστε στα νομικά λόγια και θα πρέπει να αναγνωρίσει κανείς ότι υπάρχουν διάφορα στάδια στην ενισχυμένη συνεργασία και για κάθε από αυτά τα στάδια προσπαθούμε να εντοπίσουμε σημεία συμφόρησης ε, και ε, τρόπους πρόωθησης. Αλλά εδώ θα ήθελα να τονίσω δύο σημαντικές παρατηρήσεις οι οποίες θα είναι χρήσιμες ακόμα και εάν ξεχάσουμε για λίγο ε, τις εμπειρίες μας από την ε, χρήση της ενισχυμένης συνεργασίας τα τελευταία 20 χρόνια. Έχουμε, για παράδειγμα, την, ε, την ίστατη λύση σε περίπτωση αποτυχίας της νομοθετικής διαδικασίας δηλαδή, σε περίπτωση που συζητιέται ένα νομοθέτημα για πάρα πολύ χρονικό διάστημα, η ενισχυμένη συνεργασία είναι κατά κάποιο τρόπο η ίστατη λύση. Επίσης, οι περιορισμοί ε, του, της ενισχυμένης συνεργασίας οδηγούν σε ειδικέ νομοθετικές διαδικασίες στον τομέα ε, δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Και αυτό έχει να κάνει με την ενισχυμένη ε, πλειοψηφία που χρειάζεται Και γι' αυτό υπάρχουν, για παράδειγμα, προϋποθέσεις ότι δεν θα πρέπει να υπονομεύεται η ενιαία αγορά. Θα διαπιστώσουμε ότι τα αποτελέσματα της νομικής ανάλυσης αντικατοπτρίζονται και στον πραγματικό κόσμο. Η τελευταία μου παρατήρηση στο σημείο αυτό, επειδή συζητήθηκε και στην προηγούμενη συνεδρίαση της ΑΦΚΟ και αναφέρεται και στην έκθεση Μπρόκ του 2014, Παραθέτω από την έκθεση Μπρέσο Μπρόκ, λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο να εφαρμόσει πλήρως τις διατάξεις της Συνθήκης για την ενισχυμένη συνεργασία μη δίνοντα συγκατάθεση σε καμία νέα πρόταση για ενισχυμένη συνεργασία, εκτός εάν τα κράτη, μέλη που συμμετέχουν εφαρμόσουν την ρήτρα γέφυρα, ε, το άρθρο 333 της συνθήκης, ε, να περάσουν από την ομοφωνία στην ενισχυμένη ε, πλειοψηφία. Πολλές θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επαναλαμβάνουν αυτήν την απέτηση. Η ανάλυση όχι μόνο του νομικού κειμένου αλλά και των αποφάσεων ε, του δικαστηρίου δείχνουν ότι κάτι τέτοιο οδηγεί σε περαιτέρω καθυστέρηση της διαδικασίας. Για παράδειγμα, έχουμε απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας. Ε, είχαμε την ε, νομοθεσία περί ολοκλήρωσης που ακολούθησε την απόφαση αυτή. Κάθε φορά που κάποιος γερμανός εκπρόσωπος στο Συμβούλιο συμφωνήσει για χρήση της ε, ρήτρα γέφυρας και οι δύο βουλές της Γερμανίας και το Bundestag και το Συμβούλιο ε, πρέπει να συμφωνήσουν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους ε, και αυτό βλέπουμε ότι δεν εφαρμόζεται πλήρως. Όσον αφορά τον πραγματικό κόσμο, κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στα διάφορα πλαίσια. Ε, σαφές είναι ότι έχουμε ένα χάσμα ανάμεσα στις χώρες που συμμετέχουν ε, στην Ευρωζώνη και αυτά που δεν συμμετέχουν. Έχουμε ε, για παράδειγμα και τον ε, φόρο επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών που δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Εφαρμόζεται μόνο από, την κράτος, από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και μόνο η Βουλγαρία από τα νέα κράτη-μέλη συμμετέχουν εκεί βλέπουμε ότι τα, ότι τα κράτη της Βορειοδυτικής Ευρώπης είναι πολύ πιο πιθανό να συμμετέχουν ε, στις ε, περιορισμένες συνεργασίες από ότι οι χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης και έχουμε την ε, Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σουηδία και την Πολωνία που βρίσκονται επίσης στην περιφέρεια ενώ βλέπουμε ότι ο γαλλογερμανικός άξονας είναι ε, καθοριστικός. Τα δύο μεγαλύτερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο συμμετέχουν σε όλα τα προγράμματα ενισχυμένης συνεργασίας, αλλά ήταν ε, και από τα ιδρυτικά μέλη. Κάποιες τελευταίες παρατηρήσεις από μένα, όπως ήδη είπε ο καθηγητής Βέσελς, έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο των ε, ε, τομέων ενισχυμένης συνεργασίας. Μέχρι στιγμή βλέπουμε τα εξή, ότι οι τρει από τι τεσσέρις ε, υποθέσει, υποθέτουμε ότι ο φόρο επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών είναι μισή υπόθεση ακόμα. Οι τρει από τι άλλε τέσσερι, λοιπόν, εμπίπτουν στον τομέα δικαιοσύνη και εσωτερικών. Ε, κάτι που μπορεί να εξηγηθεί από αυτή τη λειτουργία φιλτραρίσματος που σας περιέγραψα πριν. Το Κοινοβούλιο αποκλείστηκε λοιπόν ήδη από την πρώτη φάση. Μόνο σε περιπτώσεις ε, που δεν, έχουν, που δεν είδαμε ακόμα, ε, όπου χρησιμοποιείται το άρθρο 333, δεν αποκλείεται το Κοινοβούλιο. Επίσης, ε, η ιεράρχηση υποθέσεων χωρίς ε, θεσμοθέτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ε, μην ξεχνάμε ότι και ο φόρος επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών μας βρίσκει ακόμη πιο αρνητικούς από ό,τι οι εμπειρογνώμονες πέρσι είχαν πει εδώ στην Επιτροπή. Δεν βλέπουμε να υπάρχει δυνατότητα για ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Μία τελευταία παρατήρηση από μένα. Η διάρκεια της ενισχυμένης συνεργασίας πάντα εξαρτάται από το πώς την υπολογίζει κανείς, αλλά γενικά 4 με 12 χρόνια διαρκεί από την αρχική νομοθετική πράξη μέχρι την δημιουργία αυτής της υπομάδας Και αυτό θα πρέπει να το λάβει κανείς υπόψη αν θεωρεί ότι αυτή η προσέγγιση θα οδηγήσει σε μια πιο δυναμική, πιο αυθόρμητη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι, τι άλλο θα πρέπει να δούμε και πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε. Το πρώτο που έχουμε πει είναι ο κύκλος αυτής της ε, ρύθμισης. Μέχρι τις μέχρι αξιολογήσεις μας, αυτή η συνεργασία ε, δύσκολα προχωράει μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Υπάρχουν πολλές ε, δυσκολίες, μποτιλιαρίσματα, προκειμένου να προχωρούν σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό και πολλά προβλήματα λύνονται εκτός ηθικών. Ένα από τα σημεία που βλέπουμε είναι ότι πολλές χώρες προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματα και ε, κοιτούν προς κάτι, στρέφονται μάλλον προς τη λύση που θα ήταν ε, συνθήκες δορυφόροι. Ένας από τους λόγους γι' αυτό είναι ότι όλο και περισσότερο έχουμε αυτή τη διάσταση ανάμεσα στο κέντρο, που θα ήταν ας πούμε οι παλιές χώρες μέλη, τα μέλη της Ευρωζώνης, και οι περισσότερες από την άλλη χώρες ε, που προσχώρησαν στην Ευρώπη αργότερα. Αν δείτε την διαδικασία και σας συστήνω κάποια στιγμή να προσπαθήσετε να εξηγήσετε σε φοιτητέ πώς λειτουργεί ενισχυμένη συνεργασία και θα διαπιστώσετε ότι ούτε εσείς ίδια δεν καταλαβαίνετε περί τίνος ακριβώς ε, πρόκειται δεν χρειάζεται, δηλαδή δεν φτάνει να διαβάσετε το κείμενο, πρέπει πραγματικά να καθίσετε και να το μελετήσετε. Να διαβάσετε δύο και τρεις φορές το κείμενο, να καταλάβετε. Μιλάει μεν για ευελιξία, αλλά οι ρυθμίσεις οδηγούν σε πολύ μεγάλη δυσκολία να χρησιμοποιηθεί αυτή η ευελιξία. είτε πρόκειται για το περιβάλλον, είτε οι επιχειρήσεις εύκολα θα πάνε στις χώρες που έχουν χαμηλότερες προδιαγραφές. Έπειτα υπάρχουν πολιτικές που επηρεάζουν άλλες πολιτικές. Πάντα υπάρχει αυτή η αλληλεξάρτηση. Και υπάρχει και αυτή η κοινοτική ορθοδοξία. Δεν θα το έλεγα με την αρνητική έννοια, αλλά αν μη τι άλλο δυσκολεύει στην συσσόρευση κοινοτικού και εκτιμένου. Πρόκειται λοιπόν για μια πολυπλοκότητα που θα μπορούσε να ελαφρεθεί κάπως κάνοντας μικρά βηματάκια ή αλλιώς με συνταγματική αναθεώρηση. Το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να αναλάβει ρόλο και να πρωτοστατήσει στην προσπάθεια αυτή. Μέχρι τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του. Δεν μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία ενισχυμένη συνεργασίας. Πώς να χειριστεί την ενισχυμένη συνεργασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θέτει και ο εισηγητής. Δύο δυνατότητες υπάρχουν. Η μία είναι να ακολουθήσει την συνήθη πρακτική Υπάρχει μια συνήθις διαδικασία που δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των ε, ευρωβουλευτών για το κατά πόσο προέρχονται από χώρες που ακολουθούν ή όχι ενισχυμένη συνεργασία. Και το δεύτερο είναι αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουν οι ευρωβουλευτές. Δηλαδή να είναι αλλιώ για αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία, χώρες τους δηλαδή, και αλλιώ οι υπόλοιποι. Να ακολουθήσουμε δηλαδή τη δομή της ψηφοφορίας στο Συμβούλιο. Και ίσως μπορεί να βρεθεί και ένα συμβασμός και να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική επιτροπή όπου θα συμμετέχουν μόνο οι ευρωβουλευτές ή μάλλον θα ψηφίζουν, γιατί μπορούν να είναι παρόντες όλοι, αλλά θα ψηφίζουν μόνο αυτοί που προέρχονται από χώρες που ακολουθούν την ενισχυμένη ε, συνεργασία. Αλλά βέβαια την απόφαση πρέπει να την πάρει η Ολομέλεια με απόλυτη πλειοψηφία για να υπάρχει νομιμοποίηση, νομιμότητα. Αυτά προτείνω για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα που πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο θέμα. Γιατί είναι θέμα νομιμότητας και εδώ εν παρόδο να πω ότι με την νομισματική κρίση το Κοινοβούλιο αποφάσισε τι πολιτικές πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα και τι πιστώσεις θα έπρεπε να δώσουν η Ολλανδία, η Γερμανία και αυτά τα αποφάσισαν μαζί ευρωβουλευτές που έρχονταν και από την Πολωνία, τη Δανία και δεν ξέρω τι. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρόκειτο για κρίση νομιμότητας. Εδώ συμμετέχουν μόνο κάποιες χώρες στην ενισχυμένη συνεργασία, οπότε πώς μπορούν να αποφασίζουν όλοι. Αν συναποφασίσεις πρέπει να περνάνε τα μέτρα και από το εκλογικό σου σώμα. Ξέρω ότι έχουν συζητηθεί τέτοια επιχειρήματα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν είναι μαγική λύση η ενισχυμένη συνεργασία, αλλά είναι χρήσιμη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να δει ποιες θα είναι οι εσωτερικές διαδικασίες. Και τώρα έχουμε τον Αλάν, θα μιλήσετε τώρα, γιατί μετά θα μιλήσουν και οι σκιώδεις. Ε. Οι Οι η Mercedes θέλει να μιλήσει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Για την ώρα πρέπει να πω ότι άκουσα τα του ενδιαφέροντος τα όσα υπόθηκαν και έλαβα υπόψη και τις εκκλήσεις για παρέμβαση του Κοινοβουλίου. Αλλά θα σταθώ σε αυτό, διότι έχουμε καθυστερήσει πολύ και θα προτιμούσα να έχουμε το χρόνο να δούμε και το κείμενο για να το εξετάσουμε. Βέβαια το σχέδιο εκθέσεως το έχουμε και θα προβληματιστούμε δεόντως και θα συζητήσουμε το συγκητή. Δεν έχουμε μείνει πίσω. Μόνο μία ψηφοφορία έχουμε που πρέπει να κάνουμε πριν από 12.30. Έχεις τη δυνατότητα να μιλήσεις τώρα. Δεν ξέρω αν κάποιος από την ομάδα των σκιωδών θέλει να λάβει το λόγο. Ο, ο, κ. Μέσσερ Σνιτ δεν είναι εδώ. Ο Σάρς Γκέρενς δεν θέλει να μιλήσει. Χέλμουντ Σόλτ, ούτε αυτό θέλει. Είναι εδώ. Πασκάλ Ντιουράν, θε να μιλήσει. Ουχή. Ο Φάμπιο και αυτό δεν είναι εδώ. Χέροφ. Αλλά μπορεί να το κληρώσει λοιπόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω εκφραζόμενος εκ μέρους όλων των σκιωδών λέει χαριτολογώντα ο κ. Λαμασίου. Να ευχαριστήσω εκ νέου και να συγχαρώ εκ νέου την ομάδα αυτή που πραγματικά απάντησε στις τεθήσεις ερωτήσεις μας. Συμφωνούμε τις απαντήσεις τους. Πρέπει να το κουβεντιάσουμε μεταξύ μας αυτό. Ήταν ακριβώς αυτό το πνεύμα που θέλαμε να συζητήσουμε το θέμα της συνεργασίας. Λοιπόν, της ενισχυμένης συνεργασίας. Το πρώτο που διαφαίνεται σαφώς αν ήταν μακρές οι διαδικασίες, αυτό δεν οφείλεται στις ίδιες τις διαδικασίες, αλλά στην έλλειψη πολιτικής βούλησης. Απόδειξη άλλωστε αυτού, τη στιγμή που υπήρξε μεγάλη πολιτική βούληση σε ύψιστο επίπεδο στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όσον αφορά εξωτερική πολιτική, την ΠΕΣΚΟ, σε ένα χρόνο λύθηκαν τα πάντα. Όλες οι διαδικασίες λειτουργήσαν σε λιγότερο σημαντικά θέματα, πολιτικά λιγότερο σημαντικά, Έμειναν σε επίπεδο υπουργών και υψηλών αξιωματούχων τα θέματα και βλέπουμε ότι όσον αφορά τα θέματα που μέχρι τώρα οδηγούσαν σε ενισχυμένη συνεργασία ή σχέδιο ε, αυξημένη συνεργασία, δεν είχαν ε, στερνιστεί το θέμα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Υπήρχε βούληση σε ένα επίπεδο κατώτερο της Συνόδου Κορυφής που εκφραζόταν από κάποιες ε, χώρες και όχι σε άλλες. Οπότε είναι ατέρμονε οι διαδικασίε σε αυτήν την περίπτωση. Χρειαζόμαστε πολύ χρόνο να καταλήξουμε κάπου και πολύ συχνά ε, δημιουργούμε μηχανισμούς ε, περιπλοκότατου για να καταλήξουμε σε αποτελέσματα απογοητευτικά. Και όπως είπατε, κύριε καθηγητά, αυτή η διαδικασία ε, σχεδιάστηκε από τις συνθήκες για μεγαλύτερη ευελιξία, ευελιξία λοιπόν, και ταχύτητα, πολύ συχνά αποδεικνύεται πιο μακροχρόνια και περίπλοκη από την παραδοσιακή, την απλή διαδικασία. Τα καλά μαντάτα είναι ότι στα πορίσματα της μελέτης σας, αυτά που είπατε επίσης προφορικά, βλέπουμε ότι μπορούμε να, να δημιουργήσουμε κάποιο προσχέδιο που θα μπορούσαμε να προσαρμόσουμε σε διαφορετικά θέματα. Αυτό θα απαιτήσει βέβαια το ότι τα θεσμικά όργανα θα λάβουν υπόψη αυτή τη δυνατότητα, αυτή την επιλογή. Δεν είναι μαγικός τύπος. Τίποτα δεν υπάρχει μαγικό στην πολιτική άλλωστε. Ε, δεν είναι πλήρης εργαλειοθήκη, αλλά είναι από τα σημαντικά εργαλεία της εργαλειοθήκης. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενδιαφερθεί για αυτή τη δυνατότητα, να οργανωθεί ούτως ώστε να εξασφαλίσει μια παρακολούθηση και μια επέκταση τη διευρυμένη συνεργασία, ενισχυμένη συνεργασία, να οργανωθεί κατάλληλα και το Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει και το πρόβλημα που θέσατε. κάπω προκλητικά, αλλά σωστά, καλά κάνετε και το θέσατε. Δηλαδή τι είπατε, μήπως έναντι ενισχυμένη συνεργασία, όλοι οι βουλευτέ, ακόμα και εκείνοι που προέρχονται από χώρε που δεν ανήκουν στην ενισχυμένη συνεργασία, μπορούν να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Μια πτυχή του θέματος. Άλλη πτυχή θα πρέπει κατά άποψή μου το Ευρωκοινοβούλιο όταν καταλαβαίνει σε κάποιου τομεί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παρά μόνο αν στηρίξουμε τη δράση κάποιων πρωτοπόρων χωρών ελπίζοντα θα ακολουθήσουν οι άλλε, όπω το κάναμε με την Νομισματική Ένωση, όπω με το Σέγγεν όπω κατά κάποιο τρόπο το κάναμε με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο θα πρέπει να διοργανωθεί το Κοινοβούλιο να εξασφαλίζει μια συνέχεια και να μεριμνήσει ούτω ώστε η διαδικασία να καταλήξει σε αποτέλεσμα υπό καλές συνθήκες. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Άλλο σχόλιο. Πολύ ενδιαφέρον ουσιαστικά αυτό που είπατε, ότι η μόνη ενισχυμένη συνεργασία που μπορούμε να πούμε ότι πέτυχε ήταν στο διαζύγιο, για το διαζύγιο. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτή για το matrimonial property θα επιτύχει, αλλά θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Όμως, λοιπόν, είμαστε σε ένα τομέα αρμοδιοτήτων που είναι η 100% εθνική αρμοδιότης. Δυνάμει του άρθρου 91 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσης στα πλαίσια δικαστικής, διοικητικής συνεργασίας και λοιπά τι μπορούμε να κινηθούμε. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί, το λέω αυτό, διότι δια, βλέπουμε να βάλουμε υπόψη ότι τα 10 με 13 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες που σήμερα ζουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα διαφορετική από τη χώρα καταγωγής τους, βλέπουν στην καθημερινή του ζωή, στην επαγγελματική του ζωή, κοινωνική ζωή, στην οικογενειακή του ζωή, ότι υπάρχουν προβλήματα νομικά και διοικητικά ανεπίλητα. Γιατί? Διότι τα περισσότερα θέματα άπτονται του εθνικού δικαίου. Και αν θέλουμε να διευκολύνουμε τη ζωή αυτών των ανθρώπων, Έχουμε ανάγκη είτε να βρούμε λύσεις για σύγκρουση εθνικών νομοθεσιών όπως το διαζύγιο και ο χωρισμός, είτε να προτείνουμε ένα 28ο καθεστώς ε, με δυνητική εφαρμογή που μπορεί να το επιλέγει κανείς που συνάπτει μια σύμβαση που συμμετέχουν δύο-τρία κράτη γάμος, συνειδιοκτησία, ό,τι άλλο μπορεί να είναι. Και έρευνα που κάναμε στις ομόσπονδες χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως καταδεικνύει ότι στα ομοσπονδιακά συστήματα όλα τα επίπεδα κάτω από ομοσπονδιακό, τα ομόσπονδα κράτη, στη Γερμανία, οι επαρχίες, τα προβένς της Γαλλίας, τα states, οι πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ένα σύστημα συνεργασίας για να καταλήξουν σε νομοθεσίες σχεδόν κοινέ του τομείς που αφορούν την καθημερινή ζωή των πολιτών. Αν μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε τη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας με μια ερμηνεία αρκετά διευρυμένη μέσω του καταλήλου ή των καταλήλων άνθρων, των 91 κάποιο άλλο, νομίζω ότι θα είναι ένα καλό εργαλείο για τους πολίτες. Αντιστρόφως τώρα, όπως υπενθυμίσατε, το Fiscal Compact τι δείχνει και μας εκπλήσει αυτό που δείχνει, αλλά είναι και αποτελεσματικό αυτό που δείχνει. Ότι είναι αποτελεσματικό, κανείς δεν το αφισβητεί. Εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει απόφαση του ΔΕΚ αντίθετη. Ότι είναι δυνατό να περάσουμε μια δικυβερνητική συνθήκη μεταξύ κρατών, μεταξύ δορυφόρων βάσει της, του τύπου που προτείνατε, κινητοποιώντα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όπω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιήθηκε στο Fiscal Compact, όπω και το Κοινοβούλιο, το άρθρο 13 προβλέπει ότι το Δημοσιονομικό Σύμφωνο μπορεί να ελέγχεται από το Κοινοβούλιο μέσω μια συνελεύθερη διακοινοβουλευτική που συμπεριλαμβάνει μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωκοινοβουλίου. Και θεωρώ ότι είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα και αυτή. Διότι για μια ακόμη φορά, σαν θεσμικό όργανο, προτιμούμε την κοινοτική μέθοδο. Προτιμούμε τα 27 κράτη τώρα πια, 27 κράτη-μέλη, να συμμετέχουν σε όλες τις πολιτικές. Αλλά εάν είναι μια προϋπόθεση για να προχωρήσουμε και να σεβαστούμε την Ένωση στην ποικιλομορφία της, σε κάποιου τομεί για κάποιες χώρες, που μπορεί να συνδέεται ιδιαιτερότητα με την εθνική ταυτότητα και δεν θα συμμετάσχουν σε κανόνες που ε, θα τις έδαιναν με τους εταίρους τους, γιατί να τα απαγορεύσουμε. Να προσθέσω ότι υπάρχει και ένα άλλος τύπος που δεν αναφέρατε. Άλλη φόρμουλα διότι ε, δεν χρησιμοποίησαμε αυτή τη μορφή συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η φόρμουλα επιτρέπει μέσω του καναδικού ε, ομοσπονδιακού χαρακτήρα, μέσω του φιντεραλισμού του καναδικού, που πρέπει να το διερευνήσουμε αυτό, αυτό που κάνει ο Καναδάς, λόγω διεκδικήσεων του Κεμπέκ, στην περίπτωση του Καναδά. Στον Καναδά τι γίνεται. Έχουμε ομοσπονδιακούς νόμους που μπορεί κανείς να εφαρμόσει δυνητικά στη διακριτική ευχέρεια κάθε επαρχίας τη δυνατότητα να εφαρμόσει τον νόμο ή να μην τον εφαρμόσει. Προφανώς. Αν συγκρίνω με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τίθεται καν θέμα να ακολουθηθούν τις πρακτικές όσον αφορά την ενιαία αγορά, ε, θεμητό ανταγωνισμό, συνθήκες θεμητού ανταγωνισμού κλπ. Δεν μπορεί, ε, κάποια πρότυπα δεν μπορεί να εφαρμόζονται μόνο σε κάποιες χώρες ε, που θέλουν να εφαρμόσουν. Ε, θα ήταν επιλεκτικό το σύστημα έτσι. Στους τομείς που αφορούν περισσότερο την ισχυμένη συνεργασία που ουσιαστικά είναι ε, αρμοδιότητες υποστήριξης. Δεν έχουν σχέση με την ενία αγορά και όπου εκεί θα μπορούσαμε να δεχτούμε ότι υπάρχουν νομοθετικές διατάξεις διαφορετικές ακόμα και αυτές που αφορούν το δίκαιο της ενώσεως σε κάποιες χώρες. Γιατί εκεί να μην μπορούμε να διερευνήσουμε μια δυνατότητα παρόμοια. Αυτά είναι τα σχόλια, αυτές είναι οι ερωτήσεις, αυτά είναι τα θέματα που θέλω να θίξω και εν ονόματι των σκιωδών εισηγητών, ε, αυτά είχα να πω. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ. Στην προηγούμενη, προηγούμενη συνάντηση της Επιτροπής μας είχαμε και την ακρόαση με όλα τα θεσμικά όργανα που μπλέκονται στη διαδικασία. Και είχαμε συζητήσει πολύ περισσότερο για το status quo, την εξέλιξη, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερο ό,τι ήδη διαθέτουμε. Οπότε η πρότασή σας ε, έχει πολλά μαγικά στοιχεία Χρειάζεται αυτή η μαγική ιδιότητα στην πολιτική, αλλιώ πώς θα τα καταφέρναμε. Πάντως ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που είπατε, που αναφέρατε όλε αυτές τις πτυχές και θα τα χρησιμοποιήσουμε σίγουρα στην έκθεση και η αρμόδια επιτροπή επίσης. Ωραία, κλείνει έτσι η συζήτηση για αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη και σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα συνεχίζουμε και περνάμε στην ψηφοφορία. Μία έκθεση έχουμε να ψηφίσουμε. Έχουμε εδώ και τον συντάκτη της έκθεσης. Ε. Είναι εδώ ο Φάβιο. Σωστά. Α, έχουμε το χρονοδιάγραμμα όχι για την έκθεση Λαμασούρ, αλλά για την έκθεση Μπρέσο. Τον Ιανουάριο, το αργότερο το Φεβρουάριο πρέπει να ψηφίσουμε. Οπότε πρέπει να συμφωνήσετε με τη γραμματεία πώς θα προχωρήσουμε. 27 Νοεμβρίου ή αργότερα, δεν ξέρω, δείτε το με τη γραμματεία. Πρέπει να αποφασίσουμε για το χρονοδιάγραμμα, έτσι. Ναι, λέει η κυρία Μπρέσο. Έχουμε ήδη ένα κείμενο. Ε, χρειάζεται να χτενίσουμε κάποια σημεία μόνο. Πάντως, μπορούμε να αρχίσουμε στις συζητήσεις προκαταρτικά. Επί του κειμένου όποτε θέλετε. Δεν ξέρω για τη μετάφραση τι χρόνος χρειάζεται. Όχι απλώς εσείς. Να ξέρετε ότι πρέπει να δώσετε προθεσμίες και στους συναδέρφους. 27. Μπορεί, μπορείτε 27. και 22 Ιανουαρίου να ψηφίσουμε. Και αλέα και εσύ. Μπορείτε για τις 27. Συμφωνήστε με την γραμματεία για να καθορίσουμε το χρονοδιάγραμμα παρακαλώ. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στην ψηφοφορία τώρα. Για να ελέγξουμε τα μηχανήματα. Όπως είπα και σήμερα το πρωί, συμφωνήσαμε για την ε, αναβολή της ψηφοφορίας της έκθεσης του Ρίτσαρντ Κόρμπετ. Αναβλήθηκε, έτσι. Τι είπα εγώ, ακυρώθηκε. Ναι, εντάξει, ακυρώθηκε για σήμερα γιατί αναβάλλεται για κάποια άλλη στιγμή. Αλλά ναι, εντάξει, λέμε αναβάλλεται πιο σωστά. Ναι. Αλλά αν έχεις κάτι να πεις για την έκθεσή σου, πρέπει να σου δώσω το λόγο. Όχι, όχι. Για την ψηφοφορία που θα κάνουμε. Θέλω να πω στους συναδέλφους του ΕΛΚ ότι μετά από ένα εσωτερικό πραξικόπημα μέσα στο ΕΛΚ, εγώ θα ηγηθώ της ψηφοφορίας. Βέβαια αυτό το πραξικόπημα εντό εγωγικών λύγει με τη λήξη της ψηφοφορίας, έτσι. Και Φάμπιο, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να κάνω πραξικόπημα εγώ. Ήθελα απλώ να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου για την έξοχη δουλειά που έκαναν. Η συνεργασία πραγματικά ήταν πάρα πολύ σημαντική και εσά, Πρόεδρε, διότι για μερικά λεπτά μου επιτρέψατε να κάνω μια αναβολή και να μπορώ να συμμετάσχω στην ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή μα. Ακολουθήσαν παρόμοια προσέγγιση όσον αφορά το θέμα τη πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων και τη τροπολογία των συναδέλφων που είχαν ακολουθήσαν την ίδια κατεύθυνση που είχαν και δικέ τροπολογίε. Θα πρέπει λοιπόν να επιβεβαιωθεί ο ρόλο του Κοινοβουλίου, να γίνει ε, να χρησιμοποιηθούν ήδη οι πόροι, έσοδα και έξοδα ισορροπηθούν και έχουμε κοινά σημεία και τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι θεμελιώδη σημασία να εντοπίσουμε τα περιθώρια όπου η δράση σε επίπεδο ένωση δημιουργεί και δημιουργούσε μεγάλη προστιθέμενη αξία, ούτω ώστε να γίνεται προφανή η χρησιμότητα για του πολίτε ε, ε τη διακυβέρνηση. Ευχαριστώ του κοιόδη ηγητέ. Ευχαριστώ και εσά, ε, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ε, δεν έχουμε ψηφίσει ακόμα, ελέγχουμε τα μηχανήματα, έτσι. Μπορούμε να κάνουμε τη δοκιμή. Ψηφίσατε. Ωραία. Τροπολογία 43, υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροποποίηση 4. Υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Άρα τι ψηφίζουμε τώρα. Δεύτερο τμήμα. 44. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ελέγχουμε λοιπόν για το δεύτερο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. 12 υπέρ, 11 κατά. Τροποποίηση 1 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροποποίηση 2 υπέρ, κατά. απόχέ, εγκρίνεται. Τροποποίηση 3 υπέρ, κατά. απόχέ. θα ελέγξουμε για την τροποποίηση 3. Ψήφιστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. 13-9. Τώρα περνάμε στο ψήφισμα. Τροπολογία αριθμός 1 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Τροπολογία 1. Πέρας. Εγκρίθηκε. 12-11. Σύμφασμος 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Θα ελέγξουμε τροπολογία 6. Ψηφίστε. Τροπολογία 6, ναι. Τροπολογία 6, εντάξει. Πέρας. Απορρίφθηκε. 10-13. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9. Εδώ πρέπει να λέει move to, αντί για move in. Ωραία, 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Τροπολογία 10, μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας. Απορρίπτεται. Δεν σας ακούω, δεν ξέρω τι λέτε, αν διαμαρτύρεστε ή κάτι άλλο. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε τροπολογία 12. Ψηφίστε. Τέλος, απορρίφθηκε 11-12. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά, α, να ελέγξουμε 21. Συμφίστε παρακαλώ. Πέρας εγκρίθηκε. 12-11 τροπολογία 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ, θα ελέγξουμε. 30 ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. 5-18. 31 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 38. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε 10-11. Τροπολογία 39 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ονομαστική, μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας. 20 υπέρ, 3 κατά, εγκρίθηκε. Σας ευχαριστώ. Και τώρα, ολοκληρώσαμε. Θα συναντηθούμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια για το μέλλον της Ευρώπης, με επίτροπο, προεδρία και συνάδελφοι από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Οπότε, δυόμιση αρχίζουμε εδώ στην ίδια αυτή αίθουσα. Παρακαλώ, έλεξε συνεδρίαση.